Καλώς ήρθατε. Καθίστε παρακαλώ στη θέση σας. Bene. Innanzitutto bentornati a tutti. Καταρχήν σας εύχομαι καλή επάνωδο. Ελπίζω να καταφέρετε επίσης να ξεκουραστείτε από τους τριμερείς διαλόγους. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση μερισίας διάταξης. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις εγκρίνετε Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 19 η και 20 η Ιουνίου, 26 η Ιουνίου και 8ης και 9ης Ιουλίου. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ε, θα εγκριθούν στο τέλος της συνεδρίασης. Καλώς ήρθατε την κυρία Σούσανσον, νέα ε, βοηθό μας. Θα ασχοληθεί με το θέμα των υποψηφίων χωρών. και τον κύριο Φιλίπ Ποστίν του Κοινοβουλίου της Μακεδονίας, λέει ο Πρόεδρος. Ε, η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στο ίντερνετ μέσω web streaming. Στις 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες επίσης να σας ενημερώσω ότι λαμβάνει χώρα ή το συνέδριο ε, για την, τον γαλακτοκομικό τομέα ε, μετά το 2015. Είναι μια συνάντηση την οποία διοργανώνει η Επιτροπή η Επιτροπή και μας έχει προσκαλέσει. Στο τέλος της συνάντησης της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα μια κοινή συνάντηση συντονιστών με τους σκιώδεις ηγητές. Για να δούμε το πρόγραμμα σιών της Λιθουανικής Προεδρίας. Τα σημεία στα οποία έχουμε πετύχει συμφωνία με το Συμβούλιο θέματα των δημοσιονομικών προοπτικών, τα οποία δεν συμπεριλήφθησαν στις 26 Ιουνίου, στον συμβασμό της 26 Ιουνίου. Να σας ενημερώσω επίσης ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες που μιλούν τα μέλη της Επιτροπής μας. Περνάμε στο σημείο 5. Γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, όλα τα τμήματα κυρία Ταντσίλα, συγγήτρια, έχει ζητήσει το λόγο. Θα της τον δώσω αμέσως. Θα συζητήσουμε τις 21 τροπολογίες που προτείνονται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Γραμματεία για τη συνεργασία του και του συναδέλφους επίση, όλοι εκείνοι οι οποίοι συνεργάστηκαν για την έκθεση και ήθελα να σα πω ότι εγώ θα αποσύρω ε, το 15, το 19, επίσης σα ευχαριστώ. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Έχουμε μόνο 21 τροπολογίες να ψηφίσουμε. Οπότε και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε διανατάσσεως στι χειρό, Και έτσι αυτό θα εξυπηρετήσει του ανέδρους που έχουν ξεχάσει τις ε, κάρτε του την ψηφοφορία. επομένω. πάμε στην 5.307 ε, υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ε, 53.01 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5304 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-03 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53-1-4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι 3, 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53, 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53, 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53-0, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53.02 υπέρ κατά αποχές τώρα όμως θα πρέπει να κάνουμε καταμέτρηση για το 53 53.02 ψηφίζουμε ε, σηκώστε το χέρι είστε υπέρ κρατήστε το ψηλά καλώς κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται με ευρία πλειοψηφία. 53 είναι υπέρ, κατά. Συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για το 53-09. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται 53-17. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται... Συγγνώμη, αλλά παραλείψαμε μία τροπολογία. Κατά λάθο θα πρέπει επομένω να επιστρέψουμε προ τα πίσω. Να πάμε στην 53-16 και να ψηφίσουμε και εκείνη που την παραλείψαμε. 53-16 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. τελευταίε δύο τροπολογίε αποσύρονται. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Και τώρα πάμε στο σημείο 6. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό του 2014, κύριε Νταντσίλα, είναι και σε αυτή την περίπτωση η εισηγήτρια. Να δούμε το σχέδιο γνωμοδότηση. Ήδη ψήφισαμε τις τροπολογίες στις 17 Σεπτεμβρίου. Είπαμε ότι πρόκειται να συζητήσουμε το τι θα γίνει και πρόκειται επίση εκεί να τοποθετηθούμε για τις προτεραιότητές μας και για τα πιλωτικά προγράμματα και τις ε, δράσεις που έχουν προτεραιότητα. Να μην ξεχνάτε ότι οι προθεσμίες τροπολογίες ε, ορίζεται αύριο το μεσημέρι στις 3 Σεπτεμβρίου. Και τώρα. Να δώσουμε για άλλη μια φορά το λόγο στην εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο της έκθεσης περιλαμβάνει 10 σημεία και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω ότι λυπάμαι βαθύτατα και το έχω επαναλάβει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Λυπάμαι λοιπόν που ο μηχανισμός και οι εφαρμογές τους σημαίνει για τους ε, αγρότες μειώσεις περικοπές περίπου 5%. Αλλά δεδομένε της συνένεσης που έχει επιτευχθεί θα πρέπει να τους εφαρμόσουμε τους μηχανισμούς αυτούς. Επίσης θα πρέπει να τονίσω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις μη καταβληθήσεις πιστώσεις και αυτό αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να ξεκινήσουμε σωστά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 κυρίως λόγω του μειωμένου ύψους των πιστώσεων πληρωμών για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη της υπαίθρου βάσει του Αγροτικού Ταμείου θα περικοπεί κατά 5,5% σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις και αναμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελε κανείς να πάρει το λόγο για τα θέματα αυτά. Όχι. Από την Επιτροπή. Θέλει κάποιο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Διευθυντή ε, Λόγκο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Ντάντσιλα για το γεγονό ότι έδειξε ανοιχτό πνεύμα για τα, για τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαμε, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στην τελευταία μας παρουσίαση, θα ήθελα να τονίσω ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δυστυχώς αποτελεί αναγκαίο κακό, απέτηση σε ό,τι αφορά την τήρηση των ανώτατων ορίων. Και εμείς πρέπει να ορίσουμε πώς ορίζονται οι άμεσες πληρωμές και σε ό,τι αφορά τα θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ για την κατάρτιση της έκθεσης. Έχουν προσθεθεί κάποια σημεία σε ό,τι αφορά την αρχική μας πρόταση και ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τις πληρωμές για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και αν λοιπόν δεν υπάρχει κανείς άλλος που να ζητά το λόγο, να περάσουμε στο σημείο 7 της σημερινής διάταξης για τις μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη και την χρηματοδότηση, παρακολούθηση για διαχείριση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο κ. Ντες είναι ο εισηγητής, αξιότιμε συνάδελφε. Δεσμευτήκαμε προκειμένου να εφαρμοστεί αυτή η κοινή γεωργική πολιτική τον Μάιο του 2014. Παρόλα αυτά χρειάζονται μεταβατικές διατάξεις για την, ε, τον καθορισμό των τεχνικών όρων και για την συνέπεια και συνοχή σε ό,τι αφορά τα μέτρα αυτά για την ανάπτυξη της Πέτρου. Τα μέτρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να δημοσιεύονται και να δημοσιεύονται μάλιστα μέχρι τα τέλη του έτους και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχουν ψηφιστεί για να υπάρχει και περιθώριο διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο μέχρι την Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Αυτό λοιπόν θα καθορίσει και όλες τις συζητήσεις. Και τα τελευταία εκκρεμή ζητήματα που αφορούν τις μεταρρυθμίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται σε αγγίλες μέχρι 26 Ιουνίου κάποια θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να επιληθούν σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την ευελιξία μεταξύ των δύο πυλώνων είναι πάρα πολύ σημαντικά προκειμένου να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των προτάσεων. Άλμπερτ, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση αυτή είναι πάρα πολύ φύσεως και καταβάλουμε προσπάθεια ως, Ευρωπαϊκή Πολιτική, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει ολοκληρωθεί αυτή η μεταρρύθμιση το 2014. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το χρονικό πλαίσιο προκειμένου να έχουν μια ασφάλεια σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό τους οι επόμενοι οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν θα μπορέσουν ωστόσο να τεθούν όλα σε εφαρμογή το 2014, γι' αυτό και χρειαζόμαστε μεταβατικές διατάξεις και για να υπάρξει ασφάλεια σε ό,τι αφορά τα μέσα, τα ήδη υφιστάμενα για την κυνηγεργική πολιτική. Με την επιφύλαξη των, ε, της ψηφοφορίας για το θέμα της ε, τη επόμενη επόμενης δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να κοιτάξουμε θέματα για την μείωση του γραφειοκρατικού άχθους για το τέλος πρημοδότησης το 2014 τροπολογία 8 ευελιξία μεταξύ των πυλώνων και τα κρατημέλη σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούν να εναλλάσσουν τέτοια κονδύλια μεταξύ των πυλώνων, 15% στον πρώτο πυλώνα, 10% στον δεύτερο πυλώνα. Στα κράτη-μέλη των οποίων οι άμεσες πληρωμές είναι κάτω του 90% του μέσου όρου. Ύστερα, έχουμε και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση μεταξύ δύο προγραμμάτων, το οποίο είναι, τα οποία είναι το ένα μετά το άλλο. Τροπολογία 16. Ύστερα πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών για το 2016 προκειμένου να είναι δυνατή μια προετοιμασία με τη νέα αυτή η κατεύθυνση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται χρόνο για να υπάρχει ομαλή μετάβαση και να μην υπάρχουν διπλές επιδοτήσεις για το πρασίνισμα. Είναι λοιπόν σημαντικό τα θέματα που αφορούν το greening να εφαρμοστούν με ίσο και ταυτόχρονο τρόπο στα κράτη-μέλη. Για να μην παρουσιαστεί η κατάσταση που έχουμε δει στο παρελθόν, κάποιες χώρες να έχουν ολοκληρώσει την προσπάθεια και κάποιες όλες όχι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει πριν από το πέρας του έτους να ορίσουν μεταβατικές διδάξεις συγκεκριμένες που θα τροποποιούν τη σχετική νομική πράξη. Νομίζω ότι έτσι ουσιαστικά απεικονίζεται και αποτυπώνεται συναπτικά η έκθεση. Σίγουρα θα υπάρξουν τεχνικές ε, προσθήκες. Μίλησα και με κάποια κράτη-μέλη. Με προσέγγισαν αυτά δηλαδή σε περιπτώσεις που υπήρχαν συγκεκριμένες επιθυμίες. Οι Φιλανδοί για παράδειγμα είχαν ε, μια συγκεκριμένη συγκεκριμένη επιθυμία σε ό,τι αφορά τη Φιλανδία. Αλλά γενικά θεωρώ ότι με την έκθεση αυτή μπορούμε να πετύχουμε μια ομαλή μετάβαση της κοινή γεωργικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει... πιστεύω ότι μπορούν να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Ξεκινάμε την συζήτηση. Μάρτιν. Εν συντομία, Πρόεδρε. μετά από δύσκολες μεταρρυθμίσεις συμφωνήσαμε σε ό,τι αφορά την γεωργική μεταρρύθμιση και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για την έκθεση την οποία κατήρτισε εδώ ο Άλμπερτ Ντες. Το γεγονός ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει κάποια εκκρεμή ζητήματα, υπάρχουν κάποια προβλήματα στην όλη, στην όλη υπόθεση, θεωρώ όμως ότι όλα αυτά θα επιληθούν τον επόμενο μήνα, τους επόμενους μήνες. Ένα σημείο όμως ε, που ανέφερε ο Άλμπερτ να γίνει αναβολή για την πρόθεση του πρασινίσματος μέχρι το 2016. Αυτό είναι πάρα πολύ ελεύθερη ερμηνεία των όσων αποφασίσαμε για την κυνηγερική πολιτική και την μεταρρύθμιση της. Και τώρα εκ των υστέρων να ερχόμαστε να αναιρούμε αυτά που συμφωνήσαμε μετά από συμφωνία με τα κρατημέλη θεωρώ ότι είναι κάτι επικίνδυνο. Δεν είναι δυνατόν. Πολύ απλά δεν είναι δυνατό και ότι η αιτιολογία ότι όλα αυτά τα προλαβαίνουμε μέσα σε δύο έτη το 2017 θα κληθούμε να αποφασίσουμε κατά πόσο για παράδειγμα οι οικολογικές εκτάσεις θα επεκταθούν από το 4 στο 7% κοιτάξτε δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια αναβολή αυθαίρετη. Αυτό θα έθετε να αμφισβήτηση τα αποτελέσματα των τρεμερών διαλόγων. Και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Κάτι που συζητήσαμε και στη συνεδρίαση των συντονιστών σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των, της υπαίθρου. Θα θέλαμε σας παρακαλώ να υπάρξει μια παράταση σε ό,τι αφορά την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ευχαριστούμε Μάρτιν. Έρικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια παρατήρηση για την παρουσίαση την ε, δικαιολογική έκθεση ε, δεν δίδονται πολλές λεπτομέρειες ε, για, τις, για τους προσανατολισμούς που θα μας προτείνει. Πρέπει κανείς να διαβάσει τις 34 τροπολογίες και γι' αυτό θα τις σχολιάσω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη πέθρου. Σύμφωνο με την ιδέα του εισηγητή να επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα μέτρα για τις επιφανίσεις για τα ζώα αλλά να εφαρμόσουν και άλλα μέτρα σε ό,τι αφορά ιδιαίτερως τον εξυγχρονισμό, τις επενδύσεις για τον εξοπλισμό, τις υποδομές, τον εξυγχρονισμό κλπ. Υποστηρίζω αυτή την ε, πρόταση γιατί με αυτόν τον τρόπο διευρύνουμε σε όλα τα μέτρα του άξονα 2 και του άξονα 3 τις ε, ενδεχόμενες πιστώσεις που μπορούν να δοθούν. Ε, προκειμένου να καλύψουμε την διαφοροποίηση τη ζωή στην Ήπεθρο και γενικά όλε τις πτυχέ. Όμως μην ξεχνάμε και τι ενισχύσει για την εγκατάσταση νέων αγροτών, ιδιαίτερα στα κράτη-μέλη που ήδη χρησιμοποιούν τέτοιου διατάξει στο δεύτερο πυλώνα. Θα ήταν κρίμα οι διαδικασίε για την εγκατάσταση των νέων αγροτών να ε, διακοπούν ε, κατά τη διάρκεια του 2014, ενώ όλοι λέμε και συμφωνούμε ότι είναι προτεραιότητα. Θα έπρεπε να επιτρέψουμε την ανανέωση των γενεών στη γεωργία. Αυτό είναι προτεραιότητά μας. Συνεπώς, θέλω να το υπογραμμίσω. Έτσι ώστε να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα κατά τη διάρκεια του 2014. Σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις, συμφωνώ με τον εισηγητή. Πρόθεσή του είναι το συντομότερο δυνατό να αρχίσει να λειτουργεί ε, το καινούργιο σύστημα ε, ενισχύσεων. Όμως θα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε ορισμένα σημερινά μέτρα έτσι ώστε να αρχίσουμε να, εφαρμόζουμε, να, αρχίσουμε να το συντομότερο ε, τα, τους κανόνες ε, ε, εθελοντικής αποσύνδεσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την κτηνοτροφία που έχει υποστεί πλήγματα το, τους τελευταίους μήνες. Πέραν αυτά, για την τροπολογία 23 που προβλέπει από το 2014 να εφαρμόζουμε το, το πρόσθετο, ε, την πρόσθετη πρημοδότηση ε, θα ήθελα να πω ότι ε, δεν θέλουμε μια αναβολή μέχρι το 2016. Ε, διαφωνώ με αυτή την πρόταση. Διαφωνώ πλήρως με τον εισηγητή μας για αυτό το θέμα. Ε, επίσης, προβλέπονται στην έκθεση διάφορα μέτρα ευελιξίας μεταξύ των δύο πυλώνων. Ε, αυτό το είχαμε υποστηρίξει και στο παρελθόν, στον τριμερή διάλογο. Ο, από την άλλη μεριά, σε ορισμένα θυμία, σημεία, ο εισηγητής ε, ε έχει ξεπεράσει την θέση του Κοινοβουλίου. Ε, για παράδειγμα αμφισβητεί την μονιμότητα των μέτρων ευελιξίας που έχουν πάρει ήδη ορισμένα κράτη-μέλη. Το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά είναι ε, προσωρινά και μεταβατικά δεν θα πρέπει να αμφισβητεί τις συμφωνίες που έχουμε καταλήξει για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Ε, Ελίζαμπετ και μετά η Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Άλμπερτ για τη δουλειά που έχει κάνει σε ό,τι αφορά την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στον τομέα της ανάπτυξης της υπέτρου. Γιατί εδώ, σε ό,τι αφορά και τις άμεσες πληρωμές, θεωρώ ότι είναι τα πιο πολλά εκκρεμή ζητήματα. Καλό είναι, θεωρώ, το γεγονός ότι ο Άλμπερτ Ντες μιλά για τα παλιά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται με νέα κονδύλια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, κυρίως για τους αγρότες να υπάρχει μια βεβαιότητα, μια ασφάλεια. Ιδιαιτέρως στη χώρα μου βλέπουμε ότι αυτός ο ελληπής κρίκος ε, προκαλεί μεγάλη ανασφάλεια στους αγρότες. Γιατί Φυσικά πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός τουλάχιστον από ένα έτος πριν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει σαφήνεια, το είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ό,τι αφορά τα μέτρα που αφορούν τις εκτάσεις στον τομέα της ανάπτυξης της υπέτρου. Όλα τα προγράμματα, όλα τα μέσα τα οποία προγραμμα... Ε, ε, χρηματοδοτούνται από τέτοια προγράμματα να χρηματοδοτούνται από μέτρα τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την έκταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτά τα μέσα να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι η προώθηση των επενδύσεων. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχει αδειάσει ο δημόσιος κορβανάς και ήταν μεγάλη η προγραμματική περίοδος και πολλές λοιπόν επενδύσεις που έχουν ξεκινήσει δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τομέα της προστασίας των ζώων. Νομίζω ότι και εδώ χρειάζεται πολύ μεγάλος προγραμματισμός και θα πρέπει να εξευρεθεί μια λύση σε ό,τι αφορά το 2014. Γιατί πραγματικά μιλάμε για μια υπερβολικά μεγάλη περίοδο χωρίς χρηματοδότηση και το ίδιο ισχύει και για θέματα και μέτρα κατάρτισης γιατί σε θέματα εκτροφής και γεωργίας είναι πάρα πολλά τα προγράμματα εκπαίδευσης και αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν και στο μεταβατικό αυτό έτος και σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες να μην τους ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση πρημοδοτήσεις για παράδειγμα τέτοιων εκμεταλλεύσεων. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα μέτρα για τους νέους ε, αγρότες και αυτά θα πρέπει να συνεχίζονται να, ε, να χρηματοδοτούνται στο μεταβατικό έτος. Θα πρέπει να ακουστεί χειρά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στην τελευταία λοιπόν αυτή η φάση, την προγραμματική, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέτρα που δεν έχουν να κάνουν με τις εκτάσεις και θα πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε ότι θα συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ελίζαμπετ, Ούλριχ και μετά ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Άλμπερτ Ντες. Θα είμαι σύντομη. Θα πω δύο πράγματα, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί το greening θα πρέπει να αναβληθεί μέχρι το 2016. Τέσσερα χρόνια συζητάμε την κυνηγερική πολιτική. Όλοι ξέρουν τι πρόκειται να γίνει και όλοι είχαν χρόνο να προσαρμοστούν. Δεύτερη πρόταση που έχω να πω, μάλιστα, να υπάρξει μία μεταφορά από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα, αλλά έχω τεράστια προβλήματα για τη μεταφορά από τον δεύτερο στον πρώτο πυλώνα. Γιατί αν θέλουμε πραγματικά να ξεφρονθούμε τις άμεσες πληρωμές, Τώρα είναι η ευκαιρία μας και μην τη χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή. Είπατε, ναι, ότι είναι τεχνικής φύσεως αυτή η έκθεση, αλλά κοιτάξτε, έχει τεράστιες επιπτώσεις στην Ήπεθρο και στους αγρότες μας και νομίζω ότι το έχουμε συμφωνήσει εκ των προτέρων ότι θέλουμε τον πρώτο χρόνο το μπέρδεμα το οποίο προέκυψε σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις να το αποφύγουμε και γι' αυτό είπαμε Old System New Money, το παλιό σύστημα με νέα χρηματοδότηση. Άρα αυτή την ε, οδό θέλω να ακολουθήσουμε, αυτή την κατεύθυνση. Οι συνάδελφοι που φοβούνται ότι μπορεί στα ψηλά γράμματα να περάσει κάτι το οποίο θα ανατρέψει τις παλιές αποφάσεις ε, να τους καθησυχάσω. Πρόκειται για μεταβατικές ρυθμίσεις και το αργότερο μέσα από ένα έτος θα έχουμε επανέλθει στα αρχικά. Συμφωνημένα. Πολύ σημαντικό λοιπόν θέμα για μένα είναι η Ήπεθρος. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή που συμπεριέλαβε τα προγράμματα για το περιβάλλον, τα επενδυτικά προγράμματα, τα επενδυτικά προγράμματα για τους αγρότες, αλλά και για την Ήπεθρο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα αυτά να παραταθούν. Το τονίζω και καλό την Επιτροπή μας να το υποστηρίξει το μέτρο αυτό. Να το συνειδητοποιήσουμε ότι ιδάλλως γελιοποιούμαστε γιατί σε όλη την Ευρώπη μιλάμε για οικονομικά προγράμματα και εδώ πέρα στον τομέα αυτό, σε, αν δεν περάσουν αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις, να προκύψουν τεράστια κενά στη χρηματοδότηση, τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα στις επενδύσεις, τα οποία δεν θα μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Δεν θα μπορέσουμε να τα περάσουμε χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είμαι σύμφωνος με τον Άλμπερτ σε αυτά που λέει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιάρ, η κυρία Ρέιμερς και μετά ο Λουίς Καπούλας. Η Μπρίτα, ευχαριστώ. Η όλη συζήτηση καταδεικνύει ότι η έκθεση αυτή προκαλεί πολλούς φόβους ότι αφορά αυτά που δεν έχουν ακόμα ολοκληρωτικά συμφωνηθεί. Όντως, μια τέτοια εποχή θα πρέπει τουλάχιστον να περάσουν αυτές οι μεταγματικές ρυθμίσεις που θα μας επιτρέψουν να τα πετύχουμε αυτά με την λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία. Τι να την κάνει ο αγρότης, την απόφαση και τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής, αν αλλάζουν 20 φορές τα έντυπα, προκληθεί σύγχυση. Γιατί τώρα μας λένε ότι θα προτιμούσαν παράταση των όσων ισχύουν για να έχουν λίγο παραπάνω αέρα, να κάνουν ίσως και κανένα δυο λάθη στην αρχή. Τέτοια προγράμματα για την πρόθεση της ε, υπαίθρου. Ξέρετε, προβληματίζουν πάρα πολύ και τους δήμους, τις κοινότητες που μας ρωτούν τι θα γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει να το σκεφτούμε όλα αυτά, γιατί θα πρέπει όλα αυτά να διευκρινιστούν. Επίσης, σε θέματα συγχρηματοδότησης θα πρέπει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Αν θέλουμε οι οικονομικά προγράμματα ξέρετε, για την αντιμετώπιση της κρίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτικέ σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λουίς Καπούλας και μετά η κυρία Λουλίνγκ. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Ντες για τη δουλειά που έκανε και για την φροντίδα που έδειξε να παραμείνει προσιλωμένος ε, στην διαπραγματευτική εντολή που έχουμε για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ με μέσα από τις παρατηρήσεις ε, του ισκιώδου συγητή ε, της ομάδας μου, του ΕΡΙΚ, και να, θα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι το οποίο δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την διαπραγματευτική εντολή που έχουμε σε ε, αφορά το πρασίνισμα, την ε, εφαρμογή των μέτρων για το πρασίνισμα ε, τα οποία ο εισηγητής τοποθετεί το 2016 ενώ η διαπραγματευτική εντολή ανέφερε το 2015 το 2015 συμφωνήθηκε άλλωστε με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της ε, διαπραγμάτευσης με αυτό. Συνεπώς η πρόταση για το 2016 θα ξανά για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Λούλινγκ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αλμπερτές. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερως για την τροπολογία 4, καινούριο άρθρο 1 που έχει ως ε, στόχο να αποφευχθεί πρόσθετη και περιττή γραφειοκρατία. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη τροπολογία για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Όπως γνωρίζετε, η εξωτερική σύγκληση θα εφαρμοστεί ήδη από το 2014. Οπότε, το ποσό των ενισχύσεων 2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί μια φορά το 2014 και άλλη μια φορά το 2015 όταν αρχίσει να εφαρμόζεται και η εσωτερική σύγκληση. Για το 2014 θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε μόνο τα ποσά των ενισχύσεων και το 2015 να καθορίσουμε ένα καινου, μια καινούργια τιμή για τα δικαιώματα πληρωμών. Έτσι ώστε να μην χρειάζεται τρεις διαδοχικές χρονιές ε, να δημοσιεύουμε ε, καινούργιες τιμές ε, των δικαιωμάτων. Αυτό για να ελαφρύνουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τώρα το πώς θα το διατυπώσουμε αυτό να το δούμε μαζί. πραγματικά θα ήταν χρήσιμο να αποφύγουμε αυτή την περιττή γραφειοκρατία. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 1.1 και την, και την τροπολογία 5, μήπως θα έπρεπε να επανισάγουμε στο σύνολό του το άρθρο 20 του κανονισμού 1698 ε, δηλαδή και το δύο λατινικό για τους νέους γεωργούς. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Καλώς. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αρχική συζήτηση. Τώρα, ήρθε να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Φάντερβαρ έχει έρθει από την Επιτροπή και κατόπιν θα λάβει το λόγο ξανά ο κύριος Ντες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο της έκθεσης. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ε, έχει να προτείνει και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η πρόταση ε, καθορίζει κάποιους κανόνες μεταβατικούς για το 2014 και θα πρέπει να εγκριθεί πριν το τέλος της χρονιάς. Και επίσης κάποιε αυτές διατάξεις θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν από την αρχή της επόμενης χρονιάς, επομένως αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το στέλνει σαν σημαντικό μήνυμα και για να γίνει επομένω αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε το περιεχόμενο του κανονισμού στα αναγκαία. Δηλαδή όσον αφορά τη μετάβαση από τι ενισχύσει και το καθεστώ του που γνωρίζουμε σήμερα προ την καινούργια κατάσταση, τη νέα ε, μεταρρύθμιση που θα λεφθεί επομένω. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτό ο οργανισμό ούτε για να ε, θεσπίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να έχουν σχέση με το 2015 για τι άμεσε πληρωμέ, ούτε επίση με κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με, την μεταβατική. Που είναι αμφισβήτητα, τη μεταβατική ε, όπως ο Μητροπολίτες 26, 27 και 28 που αφορά αυτή την, ε, αυτή την, την κατανομή των πιστώσεων για την ε, Ήπεδρο για, για ε, την περίοδο μέχρι το 2020 κατανομή ένα 100 μέλος και αυτά επομένως το πρέπει να ζητηθούν όταν ολοκληρωθεί ο κανονισμός που αφορά την ανάπτυξη της Υπέθρου όπως είναι σαφές ότι η πρόταση η οποία κατέβηκε τον Απρίλιο έχει βελτιωθεί όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το οποίο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης και αυτό ιδιαιτέρως αφορά τις ε, ε, τροπολογίες 922 που αφορά την ευελιξία μεταξύ των πυλώνων και ε, επομένως κατά αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να μην πειράξουμε την πρόταση Κομισιόν, επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, κάποιε τροπολογίε που τι προσέξαμε, τι μελετήσαμε ιδιαίτερω. οπότε καταρχήν ε, είμαστε υπέρ του. Α πούμε η 16 ότι το 2014 θα πρέπει η σημερινή πρακτική όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα, δηλαδή να μεταφέρονται τα σχετικά ποσά ε, του πρώτου από τον, στον, στον δεύτερο πυλώνα. Επίσης έχουμε την ε, 24 που αφορά τον ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει ο οργανισμός, οι οργανισμοί πιστοποίησης και επίσης την τροπολογία 25 όσον αφορά την ημερομηνία τη ε, εφαρμογή ε, ορισμένων ε, διατάξεων του οριζοντίου κανονισμού στο μέλλον. όσον αφορά την ανάπτυξη τη υπαίθρου, σα υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το τι γίνεται επίση όσον αφορά το Δημοτικό Ταμείο, διότι δεν προβλέπεται να υπάρχουν κάποιε δεσμεύσει το 2014 επί τη βάση των κανόνων του σημερινού προγραμματισμού. Και επομένω, ε, τα υπόρρια αυτή του ΦΕΝΤΕΡ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις νέες πολιτικές και τους νέους στόχους. Άρα θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των νέων πόρων για τα παλαιά μέτρα μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο. Σε σχέση επίσης και με κάποιες ε, ημερομηνίες, κάποιες ενισχύσεις που αφορούν ε, την κτηνοτροφία και οπότε θα πρέπει να δούμε το αρχικό κείμενο γιατί εδώ έχουμε κάποιες διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ε, εκδοχών του κειμένου λέγει επενδύσεις στο αγγλικό κείμενο Οπότε αυτή εδώ η διεύρυνση του κειμένου θα πρέπει να περιοριστεί στην ε, ανέψη της Πέδρου, γιατί έχουμε κάποια μέτρα ε, για τον πρώτο άξονα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, νέα, ε, για τον νέο προγραμματισμό, ε, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον άξονα 3 και 4. Επίσης ενημερωτικά σας λέω ότι υπάρχει ένα έγγραφο της Επιτροπής που έχει διανεμηθεί. Εκεί υπάρχει μια σφαιρική άποψη για τα μεταβατική μέτρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου που νομίζω θα βοηθήσουν πάρα πολύ τη συζήτηση. Όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές δεν θεωρούμε ότι είναι τόσο σωστό να προωθηθούν κάποια θέματα όπως η ε, αυτά που προτείνει το τροπολογία 8 και 34 και επίσης, ε, επίσης είναι αδύνατο τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν από τεχνικής πλευράς ε, τα του πρώτου πυλώνα το 2014 και μόνος αυτό θα πρέπει να αναβληθεί για το 2015. Επίσης θα πρέπει από τώρα να προβλέψουμε για κάποια ζητήματα, να μην μπερδεύσουμε δυσκολούς των κυβερνήσεων και επίσης το, το, το, το 16 το πρασίνισμα, ακριβώς όπως είπε ο συγκεκριτής για το 23 θα πρέπει να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα γιατί έχουμε τα διαφορετικά στοιχεία ε, για τις άμεσες πληρωμές. Όλα αυτά είναι ένα σύνολο, άρα θα πρέπει να υλοποιηθούν, να τεθούν σε εφαρμογή ταυτόχρονα. Επίσης, όπως βλέπετε, από μεγάλη προσοχή στο ότι δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε γραφειοκρατία ε, για τους διάφορους εναλλασσόμενους, για τα κρατή-μέλη, για τους αγρότες. Οπότε αυτό, ξέρετε, ανέκαθεν μας απασχολούσε. Οπότε, βέβαια, αυτή η ανακοίνωση που αναφέρεται στο 1, στην τροπολογία είναι 1, επιτρέπει το, κάποιο περιθώριο, ε, κάποιες δράσεις, για να, κάποιες κινήσεις για να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Οπότε, αφού πρόκειται λοιπόν για κανονισμό μεταβατικού χαρακτήρα, υπάρχει ενημέρωση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου να γίνει επομένω με κάποια μέτρα που είναι και θεμητό η μείωση της γραφειοκρατίας. Όμως ε, αυτό θα γίνει αλλιώς και όχι στα πλαίσια του εν λόγω, του παρόντος κανονισμού. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε τώρα θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Αλμπερντές για τα τελικά του σχόλια και κατόπιν θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και τις συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συνοψίσω τα όσα ακούσαμε. Ο Μάρτιν Χόσλινγκς μίλησε για το greening, για το πρασίνισμα. Κοιτάξτε, δεν είναι δική μου εφεύρεση. Θεωρώ και μου το έχουν πει και πάρα πολλοί ειδικοί ότι θα είναι τεράστιο το έργο για την τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για να περάσουν και να εφαρμοστούν όλα αυτά τα προγράμματα το 30% για το δεύτερο πυλώνα, για τα κρατικά μέτρα. Κατά ήταν τεράστιο, υπέρογκο του έργο και οι νομομαθείς μου είπαν ότι, ότι χωρίς να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις κατά πόσον θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Αν λοιπόν είναι νομικά δυνατόν να υπάρξει αυτή η αναβολή, θα έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουμε και έτσι θα αποτραπεί μια υπερφώτωση των κρατών μελών. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο έτσι και αλλιώ να εφαρμοστεί η μεταρρύθμιση του κοινού, της κοινής γεωργικής πολιτικής. Δεν θα αλλάξουν τα ποσά. Τα ποσά θα παραμείνουν λοιπόν τα ίδια. Αυτά τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί το πρασίνισμα δεν είναι υποχρεωτικό στο 15 κράτη-μέλη. Αυτά που είπε ο συνάδελφο. Σίγουρα θα πρέπει να υποστρεχθούν οι νέοι αγρότες και συνειδητοποιώ ποια είναι η κατάσταση και στην δική μου χώρα. Υποστηρίζουμε ως τώρα τους νέους για την προώθηση των επενδύσεων και όπως είπατε μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε για αυτά που είπε η Ελίζαμπεθ. Φυσικά θα πρέπει να χρηματοδοτούνται καλά τα προγράμματα και θα πρέπει να βρούμε λύσεις προκειμένου τα προγράμματα αυτά να συνεχίσουν ομαλά να χρηματοδοτούνται. Αυτά που είπατε τώρα στην συνάδελφε για την πρώτη και τη δεύτερη πύλωνα. Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε από μόνοι μας. Σε κάποιες ε, χώρες έχει νόημα και βλέπω εδώ πέρα για παράδειγμα τον συνάδελφο Καπούλα Σάντο ή τη, στη Βουλγαρία για παράδειγμα υπάρχουν υπερβολικά πολλά κονδύλια στο δεύτερο πυλώνα και θα μπορούσε να υπάρχει τέτοια μεταφορά. Μόνο στις χώρες αυτές θεωρώ ότι υπάρχει νόημα να γίνει προσαρμογή. Και αυτό θα μας οδηγήσει σε πιο πολύ κυνηγεργική πολιτική στην Ευρώπη. Δεν φαντάζομαι φυσικά ότι σε κάποια χώρα όπου το 10% μόνο των κονδυλίων ε, είναι στο δεύτερο πυλώνα θα πρέπει να γίνει μεταφορά από τον δεύτερο πυλώνα, αλλά στη Σλοβενία για παράδειγμα που είναι 50-50 τα κονδύλια, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ο κύριος Γιάρ υποστήριξε την πρόταση, συνάδελφε Ράιμερς, σε ό,τι αφορά μπρίτα τους κοινότητες και τους δήμους, θα πρέπει να τα συζητήσουμε κύριε Καπούλα Σάντος. Δεν θέλω να προτείνω τίποτε που να μην είναι νομικά αποδεκτό. Με ενημέρωσαν ότι αυτό ήταν νομικά δυνατόν. Θα τα συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Να ευχαριστήσω την κυρία Άστριντ Λούλινγκ για την πρόταση να μην προκληθεί επιπλέον γραφειοκρατία και σε περίπτωση που είναι δυνατόν να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα τα κονδύλια και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις της και για τα λόγια της και είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε κοινέ λύσεις τις επόμενες ημέρες προς το συμφέρον των Ευρωπαίων αγροτών και ε, προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες αυτές οι μεταβατικές ρυθμίσεις και να εγγυηθούμε πραγματικά την ομαλή μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, Άλμπερτ. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Κύριε Πόλσα. Αντιπρόεδρος, έχεις δει το λόγο. Κύριε Πόλσεν, όχι. Για το επόμενο θέμα. Ωραία. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα. Το σημείο 8. Διατήρηση της παραγωγής γάλακτος σε ορεινές περιοχές, στις ε, ε μειονεκτικές περιοχές και στις από απόκεντρες περιοχές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτο Έχουμε την έκθεση Τόρφμαν. Οι συνθήκε παραγωγής γάλακτο σε αυτές τις περιοχές είναι στο επίκεντρο τη έκθεση αυτή. Δεδομένου ότι ε, το καθεστώς ποσοστώσεων λύγει το 2015 αναζητούνται μέτρα που θα μας βοηθήσουν να αποφύγουμε την απερίμωση αυτών των περιοχών και την αποφυγή επίσης αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καλωσορίζουμε και μία αντιπροσωπή από τον Μπολτσάνο της Ιταλίας που βρίσκεται εδώ μαζί μας για να ακούσει αυτή την παρουσίαση και το διάλογο. Δίνουμε το λόγο στον εισηγητή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, σας υπέβαλα αυτή την πρόταση και το σχέδιο έκθεσης. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, ξέρετε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και στις ε, ορεινές περιοχές, όπου παράγεται το 10% του γάλακτος στην Ευρώπη και επίσης έχουμε και τις μειονεκτούσες περιοχές και την παραγωγή την δική τους. Σημαντικό όμως είναι το θέμα της ποιότητας, το ανέφερε ήδη. Όντως, στις περιοχές αυτές παραγωγής, η παραγωγή γάλακτος είναι η μοναδική παραγωγή, μέθοδος παραγωγής και δεν υπάρχουν εναλλακτικέ. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η παραγωγή αυτή. Προτείνω κάποια μέσα τα οποία θεωρώ ότι είναι απαραίτητα προκειμένου η γαλακτοπαραγωγή στις ορεινέ περιοχές να υποστηριχθεί. Και θα συνεχιστούν και μετά τις ποσοστώσεις και τα μέσα αυτά που χρησιμοποιούνται. Μιλάμε για μέσα του πρώτου πυλώνα και νομίζω ότι σε ό,τι αφορά θέματα εσωτερικής συνοχής ε, και αυτά που έχουν αποφασιστεί στην κοινωνική πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν σε κράτη-μέλη για παράδειγμα υπάρχει το ιστορικό μοντέλο και το οποίο επιβαρύνει, αν θέλετε, τις χορτολιβαντικές εκτάσεις και την παραγωγή γάλακτος κατά συνέπεια στις περιοχές αυτές. Θεωρώ ότι είναι επίσης απαραίτητο όσο δεν υπάρχει εξισορρόπηση σωστή στον πρώτο πυλώνα, να υπάρχει δυνατότητα συνδεδεμένης πρημοδότησης για τα χορτοφάγα ζώα. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα στον δεύτερο πυλώνα. Η γεωργική πολιτική τα επόμενα 7 χρόνια προβλέπει συγκεκριμένα προγράμματα για συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες που καταρτίζουν τα προγράμματά τους αυτούς τους μήνες να τα καλέσουμε να λάβουν υπόψη τέτοια θέματα για την παραγωγή γάλακτος. Πολύ σημαντικό επίσης για την γαλακτοπαραγωγή στις ορεινές περιοχές είναι τα εφιστάμενα μέτρα του δεύτερου πυλώνα ή επιδοτήσεις για παράδειγμα για τις επενδύσεις. γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό κόστος, το κόστος της παραγωγής και υπάρχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Γι' αυτό λοιπόν τα κρατημέλη θα πρέπει να έχουν περιθώριο να υποστηρίξουν τέτοιες δύσκολες συνθήκες παραγωγής και εκμεταλλεύσεις τα, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιολογικής παραγωγής γάλακτος γιατί πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό της παραγωγής και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Είναι επίσης σημαντικό να υποστηριχθούν οι κοινοπραξίες στις ορεινές περιοχές. Γιατί ήθιστε στις ορεινές περιοχές να, υπάρχει, να υπάρχουν πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις και υψηλό κόστος παραγωγής κατά συνέπεια. Είναι λοιπόν σωστό και λογικό να υπάρχουν κοινοπραξίες σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την αρχολογική χρήση μηχανημάτων, εκτηρίων ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο είναι το θέμα του κόστους συλλογής του γάλακτος σε αυτές τις ε, περιοχές. Είναι, ξέρετε, μικρές, όπως είπαμε, αυτές οι εκμεταλλεύσεις και είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος μεταφοράς. Και αυτό ασφαλώς συνεπάγεται ότι το κόστος συλλογής του γάλακτος στις ορεινές και εξώχους απάκτητες περιοχές είναι ιδιαίτερα υψηλό. Και αυτό συνεπάγεται μειονεκτήματα. Θα πρέπει να υπάρξουν λοιπόν μέτρα για να αντισταθμιστεί το υψηλό κόστος συλλογής συγκριτικά με τις μονάδες σε πλέον πλεονεκτούσες περιοχές. Αυτό δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση υπέρ των ορεινών περιοχών, όχι απλά τις φέρνει στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες περιοχές. Επίσης, νομίζω ότι στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα το θέμα της εμπορίας του γάλακτος είναι πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερος επειδή έχει και τουριστική αξία. Είναι εξαρτή ψηλό το ποσοστό τουριστών στις ορεινές περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό και πραγματικά σκόπιμο να υπάρχει σωστή διάθεση στην στο εμπόριο του γάλακτος αυτού. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την επεξεργασία του γάλακτος στις ορεινές περιοχές. Πρότεινα να ακολουθεί το, ακολουθηθεί το πρότυπο της κοινή οργάνωσης αγοράς για τα απορροκυπευτικά. Και να υπάρξουν λοιπόν προγράμματα τα οποία θα υποστηρίξουν τις ενώσεις παραγωγών και στον τομέα αυτό για το θέμα, για παράδειγμα, της διείσδυσης στην αγορά, της ασφάλισης της ποιότητας, της καινοτομίας, τα προϊόντα διαφήμισης και προκειμένου να είναι, σωσ... να είναι κατανοητό γιατί αυτά τα προϊόντα γάλακτος υψηλής ποιότητας πολλούνται με υψηλότερες τιμές. Για παράδειγμα, Προσφάτως ε, εγκρίθηκε η νέα ονομασία προϊόν ορεινής παραγωγής. Και αυτό το πρόγραμμα ασφαλώ θα υποστηρίξει την ε, διάθεση και πώληση Επίσης θα πρέπει σε ό,τι αφορά το γάλα το οποίο διατίθεται στα σχολεία θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερος υπόψη το γάλα παραγωγής ναι. ορεινής περιοχής. Ίσως για παράδειγμα με κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αυτά λοιπόν πρόεδρα, σκέφτηκα σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου αυτές οι εκμεταλλεύσεις σε μειονεκτούσες, ορεινές ή απόκεντρες περιοχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις προωθήσουμε να έχουν μια ευκαιρία και αυτές μετά το 2015. Νομίζω το οφείλουμε στους παραγωγούς μας. Και ανυπομονώ να λάβω τις ε, προτάσεις των συνοδέλφων υπό μορφή τροπολογιών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν. Η αντιπρόεδρος, κυρία Πόλσεν, έχει στήσει το λόγο. Και μετά ο Ζωζέ Μποβέ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ε, Ρίκα Πάκερεν είναι η σκιώση από πλευράς ε, φιλελευθέρων. Ε, μόλις έχει γεννήσει ε, οπότε μου ζήτησε να κάνω μερικά σχόλια για την έκθεση Ντόρφμαν εκ μέρους της. Καταρχήν θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κύριο Ντόρφμαν για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Χαίρετε που η Κομισιόν και το Συμβούλιο έχουν υπογραμμίσει πως η γαλακτοκομική παραγωγή στις μειονεκτούσες και ορεινές περιοχές πρέπει να προσεχθεί διότι αυτές οι περιοχές θα υποστούν σημαντικές επιπτώσεις ε, τα επόμενα χρόνια με την λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων. Προφανώς όλος ο τομέας θα επηρεαστεί, αλλά ιδιαίτερος οι μειονεκτούσες περιοχές, ιδιαίτερος οι πιο απόκεντρες περιοχές. Η κυρία Πάκυρινεν ελπίζει ότι θα βρεθούν λύσεις προκειμένου να συνεχίσει για να συνεχιστεί η γαλακτοπαραγωγή σε αυτές τις περιοχές. Ο κύριος Ντόρφμαν εξετάζει τα προβλήματα αυτών των μειονεκτουσών και απόκεντρων περιοχών στο μέλλον. Οι περιοχές οι οποίες δεν θα μπορέσουν να προωθήσουν την ανάπτυξή τους ε, ε τόσο εύκολα όσο άλλες περιοχές. και οι ορεινές περιοχές έχουν παρόμοια προβλήματα και πρέπει να καλυφθούν. Ο κ. Ντόρφμαν προτείνει αρκετές λύσεις για το γαλακτοκομικό τομέα υπό τον δεύτερο πυλώνα με ιδιαίτερο ρόλο στις οργανώσεις των παραγωγών. Θα πρέπει όμως να προσθεθούν και κάποιες άλλες προτάσεις. Η γαλακτοπαραγωγή πρέπει, μάλλον πρέπει να δοθούν θετικά μηνύματα στους γαλακτοπαραγωγούς έτσι ώστε να τους δοθεί κουράγιο, θάρρος και υπομονή να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις τους. Η συνδεδεμένη βοήθεια ε, προτείνεται από το Συμβούλιο και, το, και την Κομισιόν. Ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση για την στήριξη των γαλακτοπαραγόνων. Όμως η κυρία Πάκερ φοβάται ότι δεν θα είναι αρκετή προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η γαλακτοπαραγωγή θα επιζήσει σε αυτές τις περιοχές. Χρειάζονται κάποια μέτρα αγοράς επίσης, δηλαδή ένα δίκτυο ασφάλειας προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις ε, τις οποίες θα υποστούν οι γαλακτοπαραγωγοί σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, χρειάζεται καλύτερη, ε, χρειάζονται ενισχύσεις για καλύτερη περιβαλλοντική προστασία. Αυτά ήθελα να πει κύριε Πάκυριν, να πω και εγώ ορισμένα πράγματα εκ μέρου μου πια. Στον βόρειο αρκτικό, στη βόρεια αρκτική περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, πολύ συχνά χρειάζεται κανείς να διατρέξει εκατοντάδες χιλιόμετρα για να βρει ε, γάλα. Ε, Ε, για την ακρίβεια για να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα από μία φάρμα στο σημείο πώληση. Ε, και αυτές οι αποστάσεις αυξάνονται. Ε, μετά, οι περιοχές αυτές είναι πολύ διαφορετικές διότι έχουν πολλές λίμνες, πολλά δάση και δεν έχουν γόνιμα εδάφη για διαφοροποίηση της παραγωγής. Συνεπώς, αν θέλουμε ε, να αλλάξουν παραγωγή ή να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες εγκαταστάσεις μεταποίησης είναι πολύ δύσκολο. Οι αποστάσεις είναι τεράστιες επίσης. Η δική μου περιοχή, για να καταλάβετε, ε, η δική μου εκλογική περιφέρεια 10.000 ε, ατόμων είναι τόσο μεγάλη όσο το Δουκάτο του Λουξεμβούργου. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί τεράστιες αποστάσεις μιλάμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στις περιοχές του βορρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζωσέμπαβε. Ζωσέμπαβε, ευχαριστούμε και Πόλσεν. Και εγώ να ευχαριστήσω ε, ε, τον εισηγητή γιατί νομίζω ότι έφεξε πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αξιοσημείωτο, αυτό το 10% που είπε σε σχέση με, τον, με την παραγωγή. Εγώ νομίζω ότι έχουμε όσον αφορά την απασχόληση 10% γιατί έχουμε εκμεταλλεύσει πολύ μικρέ και πάρα πολύ αύριο από αυτό το γάλα μεταποιείται. Οπότε και η αξιοποίηση του γάλακτο ιδίω όσον αφορά το, το, το, το, το τηρήσιο ζώνε δημιουργείται τρει-τέσσερι φορέ περισσότερε θέσει εργασία από ότι η μεταποίηση σε επίπεδο βιομηχανία. Επομένω, είναι πιο σημαντικό το θέμα πλήρω απασχόλησε. Έχουμε τη μεταποίηση, προστασία του περιβάλλοντο, ε, όλα αυτά λέγονται στην ε, έκθεση. Αυτό όμω το οποίο έχω επισημάνει ω προβληματικό δεν αφορά την έκθεση, αλλά μιλάμε για κάτι το οποίο δεν είναι στην έκθεση. Ότι όλα αυτά είναι μία συνέπεια του παραλογισμού του ότι θέλουν να σταματήσει το, το, το, το, το ζήτημα της διαχείρισης της ε, παραγωγής γιατί ακούω ε, να λένε για τις ορεινές περιοχές, τις ε, δύσκολες περιοχές. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όμως όσον αφορά τις ε, ζώνες αυτές που επιδέχονται τη βιομηχάνηση. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε την διαχείριση και γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση της παραγωγής και να μην αφήνουμε την αχαλήνωτη αγορά να το διαχειριστεί διότι πάντοτε θα υπάρχει το, το δημόσιο χρήμα για να αντισταθμίσει την καταστροφή της συγκέντρωσης της γαλακτοβιομηχανίας. Σήμερα βλέπουμε όμως την επιτάχυνση του ρυθμού αυτής της συγκέντρωσης, βλέπουμε τη βιομηχανία να εξαπλώνεται, ε, ε από 5.000 ε, ε, γαλακτοφόρες, έχουμε 50 και πάνω σε, σε ορεινές ζώνες, Επομένως θα πρέπει να επανέλθουμε και να πούμε στην έκθεση ότι θέλουμε το 2015 να ξαναέχουμε κάποιες προσθέσεις γάλακτος. Πρώτον αυτό και δεύτερον θα πρέπει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να συνεχίσουμε το έργο αυτό το οποίο ξεκίνησε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης της ε, ΚΑΠ με το Μισελ Νταντέν και θα πρέπει μένως να ενισχύσουμε την δυνατότητα να έχουμε σε κοσμένες περιοχές, στις ζώνες ε, ε, ονομασίας για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τον όγκο της παραγωγής σε σχέση με τη θέση σε εμπορία και αυτό να γίνεται με διαπραγμάτευση επί της τιμής μεταξύ των ε, παραγωγών και των μεταπηδών τόσο ώστε όλα αυτά να είναι ένα λογικό σύνολο και όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε όμως νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτά τον οποίο γινόμαστε σήμερα μάρτυρες είναι η συνέπεια μιας ιδεολογίας ε, ότι δηλαδή όλα θα τα ρυθμίσει η αγορά. Όμως αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Γεωργία. Ε, μπορεί μερικοί να στεναχωριούνται ή να χαίρονται, αλλά πάντως η ε, πραγματικότητα είναι αυτή ο πρόεδρος. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Χοφμαν, τον κύριο Ντόρφμαν για, ε, για την, το έργο του. Ε, επισκέφτηκε επισκέφθηκε πολλές ε, ορεινές περιοχές, είδε από κοντά την κατάσταση. τα προβλήματα των ορεινών περιοχών συνδέονται καταρχήν με το περιβάλλον που περιορίζει τις δυνατότητε του ανθρώπου και αυξάνει τα κόστη. Το κλίμα, οι κλιματολογικές συνθήκες επίσης αυξάνουν το κόστος, γιατί για παράδειγμα οι ταράσεις των κτηρίων πρέπει να αντέχουν πιο ισχυρές για να αντέχουν το χιόνι, για παράδειγμα λέω. Ε, θα ήθελα όμως να επιμείνω στο θέμα της απομόνωσης. Η απομόνωση στις ορεινές περιοχές, όπως αναφέρθηκε και για το βορρά της Ευρώπης, ε, η απομόνωση δεν αυξάνει απλώς τα κόστη. Ε, είναι και πηγή εγκατάλειψης, είναι και ε, αιτία εγκατάλειψης των περιοχών αυτών από τον πληθυσμό τους. Θα πρέπει λοιπόν να, δοθεί, να δίδεται στα προϊόντα μια προσθέμενη αξία επιτόπου. Όμως πολύ συχνά είναι δύσκολο να διατηρηθούν οι οικονομικοί αυτοί παράγοντες που θα επέτρεπαν έστω και μια ελάχιστη ισορροπία. Και η μεταποίηση, ναι εντάξει, καμιά φορά είναι λύση. Ε, αλλά ε, η πραγματικότητα είναι αδύρυτη. Η μεταποίηση απαιτεί πολλή δουλειά. Πρέπει καταρχήν κάποιος να παράγει το γάλα και μετά να το μεταποιεί, να του προσθέτει αξία είναι μια άλλη δουλειά, μια δεύτερη δουλειά. Οπότε αυτό που ε, φαίνεται να είναι καλή λύση ε, έχει προβλήματα. Για το θέμα λοιπόν του γάλακτος στις ορεινές περιοχές ε, έχουμε ένα γόρδιο δεσμό. Ε, ποιος είναι ο ρόλος μας, να διαπιστώσουμε το τι συμβαίνει και απλώς να κάνουμε μικροδιορθώσεις ή να θέσουμε στη διάθεση των παραγωγών πραγματικά εργαλεία για να τους βοηθήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν που δέχτηκε αυτή την, πρωτοβουλία, ε, την της πρωτοβουλίας γιατί μετά τη δουλειά που κάναμε για το πακέτο γάλακτος που είχαμε υπογραμμίσει ε, τα προβλήματα των ορεινών περιοχών ε, που όμως δεν έδωσε αποτελέσματα διότι το Συμβούλιο μπλοκάρισε το θέμα στις κοινή οργάνωση αγορών ε, θα ήταν χρήσιμο αυτή η έκθεση να υιοθετηθεί με μεγάλη πλειοψηφία ή με ομοφωνία έτσι ώστε να δώσουμε στην Κομισιόν ε, την δυνατότητα να κάνει προτάσεις και στο, κοινοβούλιο, το, και στο Συμβούλιο να συμφωνήσει μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Τα επιχειρηματά είναι πολύ σημαντικά. Κύριο Σάλβες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόρφμαν. Είναι πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση. Ήρθε στη σωστή στιγμή. Και ως και ως ηγητής ε, της ομάδας των Σοσιαλιστών ελπίζω θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του. Εγώ προέρχομαι από μια ορεινή περιοχή Μάλλον εγώ προέρχομαι από μια ε, άκρος ε, ε απομακρυσμένη περιοχή και ο ίδιο προέρχεται από μια ορεινή περιοχή, συνεπώς συνδυαζόμαστε καλά. Από την αρχή ε, θητεία μα μας ε, έχουμε εκφράσει σημαντικέ ανησυχίες για την του συστήματο γαλακτοκομικών ποσοστώσεων. Γιατί δεν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί που θα ρυθμίζουν την ε, προσφορά σε αυτόν τον τομέα. Δεδομένου ότι αυτό το τομέας έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εγώ προέρχομαι από μια περιφερειακή ε, χώρα και από μια ε, άκρος απομακρυσμένη ε, εξόχως απόκεντρη περιοχή. Οπότε γνωρίζω πολύ καλά το θέμα. Με, ανησυχεί, με ανησυχούν ιδιαίτερως οι επιπτώσεις αυτής της κατάρρησης στις άκρους απόκεντρες και τις ορεινές περιοχές που αποτελούν αντικείμενο αυτής της έκθεσης. Η γαλακτοκομική παραγωγή σε τέτοιες περιοχές δεν μπορεί να υποκατασταθεί ε, είναι η βασική ατμομηχανή των οικονομιών τους, ε, της ε, κοινωνικής συνοχής τους, τους της προστασίας του περιβάλλοντος, ακόμα και της προστασίας του, της ίδιας της επικράτειάς τους. ο εισηγητής ήρθε στις Αζόρες και είδε ότι εκεί παράγεται το 33% της συνολικής παραγωγής γάλακτος της χώρας μου. Ε, μια, επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, υποβάλει ε, έκθεση σύντομα για το θέμα της κατάργησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και πριν από ένα χρόνο εγώ συναντήθηκα με τον κύριο Τσιόλος και του έθεσα το θέμα των υπόκεντρων και των ορεινών περιοχών. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα συστήματα και ποιε είναι οι περιοχέ που υπάρχουν, που παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να εξισορροπήσουμε την οικονομική διάσταση και την ε, εδαφική διάσταση τη παραγωγή του γάλακτο. Πώ μπορούμε να διατηρήσουμε την συνεισφορά του γαλακτοκομικού τομέα στην επιβίωση των τοπικών κοινωνιών, διότι πραγματικά σε πολλές κοινωνίε είναι απολύτως απαραίτητο αυτός ο κλάδος. Ε, ο κύριος Επίτροπος θα συμπέρανε όλα αυτά στην ε, έκθεση και έχει δεσμευθεί να ξεκινώντας με την, ε, το συνέδριο της 24ης Σεπτεμβρίου έχει λέω δεσμευθεί να εξεταστεί το θέμα και εκεί στις 24 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν τα πορίσματα της μελέτης η, τάση είναι να αντικατασταθούν τα σημερινά μέτρα με τα μέτρα του πακέτου γάλακτος, αλλά κατά την άποψή μας αυτό δεν είναι επαρκές. Αυτές οι ανησυχίες άλλωστε ακούγονται και σε άλλους τομείς. Μάλλον ακούγονται σε όλη την Ευρώπη ε, από τους παραγωγούς γάλακτος. Λυπάμαι που στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ δεν ελήφθη τίποτα παραπάνω, ε, υπόψη τίποτα παραπάνω από αυτό που είχε ληφθεί υπόψη στο πακέτο γάλακτος. Δεν, λαμβάνουν μέτρα για την, δεν λαμβάνονται μέτρα για την ε, ρύθμιση της ε, ε, προσφοράς. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τώρα με αυτή την έκθεση προσφέρουμε κάτι παραπάνω και δίνουμε μια ελπίδα στους γαλακτοπαραγούς, ιδιαίτερα των πιο μειονεκτουσών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα σχόλιο θα ήθελα τώρα να κάνω. Θα ήταν χρήσιμο ε, το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης να, λαμβάνει, να λάβει υπόψη την έκθεση της Κομισιόν ε, και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει στις 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες ε, στο συνέδριο που οργανώνει ο Επιτροπός Τσιόλος. Εκεί πιστεύω ότι όσα θα ακουστούν θα ε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεσή μας. Πιστεύω λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα για τις τροπολογίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συνέδριο της 24ης Σεπτεμβρίου. Τώρα για το περιεχόμενο. Ε, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να γίνει μια θετική διάκριση που θα λαμβάνει υπόψη το σενάριο μετά την καταργήση των ποσοστώσεων στις ε, μειονεκτούσες περιοχές που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την γαλακτοπαραγωγή. Αυτή η θετική διάκριση θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραλαμβάνω, αλλά και σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηρίξουν με ιδιαίτερο τρόπο αυτές τις περιοχές για να αντιμετωπίσουν αυτές οι περιοχές την καινούρια πραγματικότητα. Με αυτό τον στόχο θα εργαστώ επί αυτής της έκθεσης προκειμένου να οθήσουμε και τα κρατημέλη και την Κομισιόν προς αυτήν την κατεύθυνση και παρακαλώ να ληφθούν υπόψη τα πορίσματα της μελέτης που θα, που θα παρουσιαστεί στις 24 Σεπτεμβρίου. Πρόεδρος, ε, Πατράου Νέβες. Έχουμε 7 ακόμα μιλτές. Κυρία Πατράου Θα ήθελα να ξεκινήσω υπογραμμίζοντας την σημασία αυτής της έκθεσης. Και από πλευράς μορφής και από πλευράς περιεχομένου. Σε ό,τι αφορά τη μορφή της. Είναι μαρτυρία ότι, για το ότι ο γαλακτοκομικό τομέας είναι σημαντικός στην Ευρώπη. Και παρόλα τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στην Επιτροπή Γεωργίας από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικός αυτός το μέσο στην Ευρώπη ε, και τον υπερασπιζόμαστε. Η λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων αποτελεί πρόκληση ιδιαίτερα για τις μειονεκτούς περιοχές. Ε, ο χρόνος για να βρούμε λύσεις ε, λιγοστεύει η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ δεν μας βοήθησε. Και τώρα αναλαμβάνουμε αυτή την γνωμοδότηση πρωτοβουλίας ακριβώς για να δείξουμε ότι ο τομέας αυτός μας απασχολεί και αναζητούμε αποτελεσματικές λύσεις. Ε, αυτά σε ό,τι αφορά τη συμβολική αξία της έκθεσης. Τώρα, από πλευράς περιεχομένου. Διαβάζοντας την εξαιρετική έκθεση ε, του κ. Ντόρφμαν, τον οποίο θέλω να συγχαρώ και δημοσίως, ε, μας δημιουργείται η σιγουριά, επιβεβαιώνομαστε στο ότι η γεωργία είναι πολύ σημαντική σε όλη την Ευρώπη, αλλά ιδιαίτερο στις μειονεκτούσε περιοχές. Είναι μια σημασία που ξεπερνάει τους οικονομικούς παράγοντες. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τη γεωργία μόνο από το οικονομίστικο πρίσμα, μόνο μέσα από το οικονομιστικό πρίσμα. Η γεωργία είναι θεμελιώδου σημασία για την Ευρώπη, για την κοινωνία των πολιτών. Εμείς είμαστε μια κοινωνία πολιτών και όχι μια αγορά. Θα πρέπει να αντιληφθούμε την κοινωνική πτυχή όλων των τομέων και αυτή η έκθεση το υπογραμμίζει ε, προβάλλει αυτή την κοινωνική διάσταση υπεράνω των οικονομικών επιχειρημάτων με τη λήξη του καθεστώτος των ποσοστώσεων και με την παρουσίαση του πακέτου γάλακτος ε, δεν θα λείψει. Ε, μπορεί να λείψει το γάλα από την Ευρώπη. Μάλιστα μπορεί να δούμε περιοχές που για δεκαετίες ή και για αιώνες παρήγαγαν γάλα να σταματήσουν να παράγουν. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση, το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να καταδικαστούν σε θάνατο ορισμένες από αυτές τις περιοχές και η Ευρώπη να μην χωρίς γάλα. Μιλάμε για μειονεκτούς περιοχές, ορεινές περιοχές, ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Η έκθεση απαιτεί αυτές οι περιοχές να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν γάλα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αντιληφθούμε τις ιδιαιτερότητές τους και να υιοθετήσουμε επαρκή και κατάλληλα μέτρα που να προσαρμόζονται σε αυτές τις ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεπεράσουμε τα οικονομικά επιχειρήματα και να σταθμίσουμε και τον κοινωνικό παράγοντα, έτσι ώστε αυτές οι περιοχές να συνεχίσουν να παράγουν γάλα. Ο εισηγητής το λέει πολύ σαφώς, εντοπίζει με μεγάλη ακρίβεια τα προβλήματα και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Μπορούν να βελτιωθούν, μπορούν να συμπληρωθούν, σίγουρα. Θα το κάνουμε μέσω τροπολογιών αλλά έλεγα ότι πέραν της, του εντοπισμού των προβλημάτων και των προτάσεων μέτρων αναφέρει καθαρά πως η παραγωγή γάλακτος ξεπερνάει το γάλα. Ε, έχει σχέση με τον τουρισμό, με την ε, προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος κλπ. Και όλα αυτά θα πρέπει να σταθμιστούν. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις υποστηρίζω τα του εισηγητή Πιστεύω ότι πρέπει να συμπληρωθούν με κάποιες άλλες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξόχους απόγεντες περιοχές, διότι ε, ο εισηγητή έχει λίγο, δείξει λίγο μεγαλύτερη ε, ευαισθησία σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των ορεινών περιοχών, ακριβώ διότι προέρχεται από μια τέτοια περιοχή. Ε, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα μέτρα αυτά λίγο πιο προσαρμοσμένα στις απόκεντρε περιοχέ. περιοχές. Ε, μην ξεχνάμε ότι οι απόκεντρε περιοχέ περιοχές είναι κατακαιρματισμένε γεωγραφικά και έχουν προβλήματα διαφορετικά από αυτά των ορεινών περιοχών. Για παράδειγμα, πολλά προβλήματα μεταφορών. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, αλλά και σε ό,τι αφορά την μεταπίση και την εμπορία του γάλατος. Θα συνεργαστώ λοιπόν πρόθυμα και με όλη μου την καρδιά με τον εισηγητή. Το έγγραφο είναι ήδη έξοχο, μας διευκολύνει και θα ελπίζω θα μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις στο πρόβλημα το οποίο όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά. Ευχαριστώ. το e Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόρφμαν και κύριε Ντόρφμαν θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μισελ Ταντάν που έκαλε τους πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και θεωρώ κύριε Ντόρφμαν ότι ακολουθείται επάξια του, το έργο του Μισελ. Όλα αυτά είναι σημαντικά σε ό,τι αφορά την συνέχιση του έργου του Μισελ και πραγματικά είναι εξαιρετική η έκθεση που προετοιμάσατε. Έχει γίνει μια ευρεία συζήτηση για το θέμα αυτό και, και η συζήτηση αυτή ακριβώς αποτυπώνει την σπουδαιότητα του ζητήματος. λέμε ότι θέλουμε ως βουλευτές θέλουμε να ακολουθήσουμε την αγορά, αλλά θέλουμε να υπάρχει και κοινωνική ευθύνη σε ό,τι αφορά το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό κύριε Τόρφμαν, και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το στείλουμε ως μήνυμα προς τα έξω. Μας ρωτάει ο κόσμος στις ορεινές περιοχές τι κάνετε εσείς για μας στις ορεινές περιοχές, στις ε, απόκεντρες περιοχές, στις μειονεκτούσες περιοχές. Η περιφερειακή παραγωγή στις περιοχές αυτές θα πρέπει να αποτελεί στόχο μας. Και αυτά συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση Dorfman, πώς μπορούμε να κάνουμε παραγωγή, μεταποίηση στις περιοχές αυτές. Για να μπορέσει ο κόσμος να συνεχίσει να ζει στις περιοχές αυτές, εάν το θέλει. γιατί στην περίπτωση αυτή μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τουριστικά τις περιοχές αυτές. Και αν κάτσουμε με τα χέρα σταυρωμένα και φύγει η χαλακτοπαραγωγή από τα μέρη αυτή, θα φύγει και ο κόσμος. Δεν είναι, ξέρετε, απίθανο το σενάριο αυτό. Είτε μιλάμε για τις Άλπεις, είτε μιλάμε για κάποιες περιοχές της Ισπανίας ή άλλες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη είναι δική μας και θα πρέπει λοιπόν να την αναλάβουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την έκθεσή σας αυτή που καταδεικνύει την ευθύνη μας για το περιφερειακό αυτό επίπεδο. Χρειάζεται κατεπηγόντως λοιπόν μια σχετική απόφαση ή δυνατόν και με μειοφωνία. Αυτό θα είναι πολύ καλό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ιδιαίτερα και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προς το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Κώστιγκεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον Herbert Dorfman για την πρωτοβουλία, για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, το οποίο αγγίζει πραγματικά πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη όπως το είπε και η κυρία Γέγκλε, όσοι ζουν και εργάζονται στις περιοχές αυτές πραγματικά ελπίζουν να βρούμε τις απαντήσεις τις οποίες έχει αφήσει ουσιαστικά, ουσιαστικά ανοιχτά, ανοιχτές ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την σχετική ε, έκθεση για το γάλα. θα πρέπει να ξέρουμε ότι το 60% των ορεινών περιοχών διατίθεται για την παραγωγή γάλακτος. Ουσιαστικά λοιπόν οι αγρότες, οι εκτροφείς στις περιοχές αυτές δεν έχουν άλλη εναλλακτική πέρα από την παραγωγή γάλακτος. Η μοναδική άλλη εναλλακτική λύση είναι η αστιφλία. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναχαιτιστεί αυτό το κύμα αστιφιλίας, να ληφθούν μέτρα τα οποία να εφαρμοστούν επιτυχώς. Είμαι βέβαιη ότι η γαλακτοπαραγωγή στην περιοχή αυτή θα διατηρηθεί μόνο εάν υπάρξουν κίνητρα. Ο κύριος Ντόρφμαν προτείνει κάποια στοιχεία, τα υποστηρίζω ανεπιφύλακτα, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι η γαλακτοπαραγωγή αποτελεί τμήμα της ταυτότητας του κόσμου στις περιοχές αυτές. Και νομίζω ότι κάτι που δεν λαμβάνουμε υπόψη σε αυτή τη συζήτηση είναι το εξή. Δεν μιλάμε μόνο για την παραγωγή αυτή, αλλά για την ε, πολύ κλειστή και πολύ αποτελεσματική παραγωγή στις περιοχές αυτές. Δεν μιλάμε εδώ λοιπόν μόνο για κάποιες περιορισμένες εκμεταλλεύσεις στην τελική ανάλυση. Και επίσης ότι για τις περιοχές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικός ο πλάτος του τουρισμού. Καμία κοινότητα, κανένας δήμος δεν μπορεί να δώσει αυτό το κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς. Αυτό το κάνουν οι αγρότες, οι εκτροφείς και το είπε η κυρία Μπάουσεν. Ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα είναι το θέμα της μεταφοράς. Πώς θα μπορέσουν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται αυτές οι μεγάλες μεταφορές, οι μακριές μεταφορές και στο μέλλον. Στην Αυστρία, για παράδειγμα, έχουμε περιφέρειες όπου πριν από 20 χρόνια υπήρχαν 30 παραγωγοί γάλακτος, πλέον είναι μόνο 3. Και άρα δεν αξίζει τον κόπο να γίνονται μεταφορές. Ποιο λοιπόν επιβαρύνεται με το κόστο αυτό. Αλλά αν δεν συνεχίσουν οι μεταφορέ γάλακτο, πολύ απλά θα σταματήσει και η παραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν είναι δικό μα καθήκον να βρούμε λύσει στα ερωτήματα αυτά. Και νομίζω ότι ο Μισελ Ταντάνα έκανε τη σωστή ερώτηση. Τι αξίζει για μας το γάλα από τις περιοχές αυτές. Δεν είναι μόνο για οικονομικό, δεν πρόκειται μόνο για οικονομικό ζήτημα, ξέρετε. Νομίζω ότι είναι πολιτικό ζήτημα αυτό, καταρχάς. Και ναι, νομίζω ότι η απάντηση είναι καταφατική. Αξίζει η παραγωγή γάλακτος σε αυτές τις δύσκολες περιοχές, τις απόκεντρες περιοχές, τις ορεινές περιοχές. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντική η παραγωγή γάλακτος και ελπίζω λοιπόν να λάβει υποστήριξη η, παραγωγή, η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Herbert Dorfman για την αξιολογική εκθεσή του. Οπότε εμείς με τη σειρά μας τώρα, είμαστε ενώπιον των πολιτικών ευθυνών μας. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι, γαλακτοπαραγωγοί παντού, να είναι κοντά στις ε, αγορές, ε, και έτσι ε, να μπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους και θα πρέπει εδώ να δούμε τι θα γίνει στις ε, ζώνες τις μειονεκτικές, τι γίνεται στις περιοχές της απότερης περιφέρειας, τις αξόχους από εκείνες περιοχές και να δούμε τι θα γίνει με την κατάργηση των προσθέσεων της 2015 επίσης. Έχουμε και το θέμα του ελευθέρου ανταγωνισμού, όπως αναφέρθηκε. Δεν είναι δυνατόν αυτό μόνο του να ρυθμίσει το πρόβλημα των μειονεκτικών και των ορεινών περιοχών. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε τι είδους οικονομίας, τι είδους δραστηριότητα μπορεί να επιβιώσει σε τέτοιου είδους εδάφη. Οπότε επ' αυτού και εμείς ερχόμαστε τώρα να λάβουμε τις ευθύνες μας και να λάβουμε υπόψη τον άνισο χαρακτήρα ε, των εδαφών και να προσπαθήσουμε να μην κάνουμε την ε, αγροτική πολιτική ακόμα πιο άνηση. Να μην ε, ανακατεύουμε τις περιοχές με τα ίδια για όλους. Αυτό θα πρέπει να πει η έκθεση. Οπότε έχουμε αυτές τις μηνευτικές περιοχές, εκεί, εκεί που υπάρχει πάρα πολύ αραιή ε, τοποθέτηση των εκμεταλλεύσεων και των ζώων, θα πρέπει να δούμε πώς, εάν τις διατηρήσουμε αυτές τις εκμεταλλεύσεις, αυτό να πτήσει την ύπεθρο γιατί υπάρχουν και θέματα πέραν της γαλακτοπαραγωγής. Είναι θέματα των ε, αποβλήτων, ε, των νερών, του, του υδατός κλπ. Οπότε όλα αυτά, όπως είπαν διάφοροι προλήσεις, πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Και έτσι θα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πολύ ευρύτερη της έκθεσης. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό μεταξύ άλλων να δούμε πώς θα υπάρχει ε, περισσότερη πρόσβαση στις ενισχύσεις του δεύτερου πυλώνα και επίσης αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε όσον αφορά τις ε, επενδύσεις και την καινοτομία. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι πιστώσεις για έρευνα και καινοτομία θα πρέπει να προσαρμοστούν στην διαφοροποίηση των προϊόντων. Γιατί εδώ μιλούμε για το γάλα. Όμως la réforme qui est en cours. Και να δούμε τι θα γίνει και με τη χειροτροφία σε αυτέ τι περιοχέ να δούμε πώ θα μπορούμε να βοηθήσουμε του παραγωγού ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τι ιδιορυθμίες των προϊόντων που σε αυτέ τι ιδιαίτερε περιοχέ ε, αναπτύσσονται. Οπότε και να, να λάβουμε υπόψη του την πολυπλοκότητα τη οικονομία σε αυτού του κλειστά εδάφια. Ε, ευχαριστώ, Ερικ, ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρώτα πρώτα. Να σας πω ότι άκουσα κάτι από τον κύριο Καπούλας Σάντος όταν ανέφερε ότι θα πρέπει να προβούμε στη σωστή διαχείριση των μειονεκτικών περιχών αλλά από την άλλη μετιά προτιμά αυτό να το κάνει με ενίσχυση χθες εξ αρχής και όχι εκ των ε, υστέρων παρέμβαση όταν πια έχει περιμωθεί η συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό λοιπόν ισχύει όσον αφορά την γαλακτοπαραγωγή. Θα πρέπει να φροντίσουμε η γαλακτοπαραγωγοί να μένουν σε αυτές τις περιοχές, να τους δώσουμε κάποια κίνητρα για να μείνουν εκεί. Το γάλα, όπως όλοι γνωρίζουμε, εκεί είναι καλύτερες ποιότητες. Και αυτό να ληφθεί υπόψη. Θα πρέπει φυσικά και το περιβάλλον να προστατευτεί όπως πρέπει. Έχουμε αυτές τις λιβαδικές εκτάσεις που κάποτε τις είχαμε για να βοσκούν τα βοηδή. Ε, όμω όμως ε, δεν χρησιμοποιηθεί αυτό το λόγο. Να, πώς εξαφανίζεται από τις περιοχές εκείνες και η χλωρίδα και η πανίδα λόγω αυτών των μεταβολών. Διότι υπάρχουν και κάποιες περιοχές όπου η φύση έχει ανακτήσει κάποιες ζώνες, κάποιες περιοχές. Οπότε, βέβαια αυτό είναι πρόβλημα ε, και στους γαλακτοπαραγωγούς και στους κτηνοτρόφους γιατί ας πούμε ε, στις αυτές τις λιβαδικές εκθάσεις, στους βοσκοτόπους έχουν επιστρέψει τα ελάφια. Οπότε δεν θα τους εγκαταλείψουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε να μείνουν εκεί αυτή η αυτοπαραγωγή, αυτή η κτηνοτρόφια, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν για να το καταφέρουμε αυτό. Μάρτιν Χόισλινγκ. Ναι, νομίζω ότι συμφωνώ με πολλά από αυτά που ακούσαμε. Έχω όμως ε, να πω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι θα ήταν καταστροφή να καταργηθεί η παραγωγή μιας περιθωριακής ε, ποσότητας. Είπε και ο κύριος Δόρφμαν ότι μιλάμε για μια στρέβλωση που μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Η διόρθωση μέσω του δεύτερου πυλώνα θεωρώ ότι είναι μια φρούτα ελπίδα γιατί ιδιαίτερος ε, σε ό,τι αφορά το δεύτερο πυλώνα τα κράτη-μέλη υπόκεινται τις πιο μεγάλες περικοπές. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για να διατηρηθεί η παραγωγή γάλακτος σε αυτές τις περιοχές και από πού θα έρθουν τα χρήματα αυτά. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα των ορεινών περιοχών. Πολλά θέματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Ντόρφμαν είναι θέματα που πλήττουν τις μικρές επιχειρήσεις που δεν μπόρεσαν, για παράδειγμα, να μετατραπούν σε εκμεταλλεύσεις παραγωγής δημητριακών και έτσι αναγκαστικά στράφονται στο γάλα. Μπορεί να πρόκειται για εκμεταλλεύσεις που είναι πάρα πολύ μικρές, δεν παράγουν αρκετό γάλα και γι' αυτό δεν αξίζει τον κόπο τελικά. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να σκεφτούμε και να βήμα παραπέρα. Μήπως αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και στην διάσκεψη της 24 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρω πώς μπορεί να διορθωθεί λοιπόν η κατάσταση αυτή σε πολλές περιοχές, αλλά σε κάθε περίπτωση Το Νότιο Τυρόλο, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα επιβιώσει όλη αυτή η περιοχή χωρίς την παραγωγή γάλακτος. Μιλάμε για κάτι το ζωτικό για την επιβίωση της περιοχής. Πολλά σωστά σημεία αναφέρθηκαν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει επί της αρχής να συζητήσουμε τη διαμόρφωση της αγοράς, να δούμε κατά πόσον θα κινηθούμε προς την απελευθέρωση τη αγορά το οποίο πραγματικά θα βλάψει τον κλάδο αυτό. Είναι αναπόφευκτο. Κύριε Σιρίτσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και, τα, και η εισαγωγή του παρουσίαση του εισηγητή και η συζήτηση αποδεικνύουν ότι το θέμα είναι ιδιαίτερα ακαθόδες. Βέβαια, εκ πρώτη όψεω ε, θα μπορούσε κανεί να πει ότι είναι απλό. Διότι πώ μπορεί να διατηρηθεί η παραγωγή σε ορεινέ περιοχέ και σε εξόχω απόκεντρε ε, περιοχές, ιδιαίτερα στο βορρά. Ε, το ερώτημα δεν αφορά μόνο την παραγωγή του γάλατος, αλλά και οποιαδήποτε άλλη παραγωγή. Το ερώτημα είναι αν πράγματι θέλουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή εκεί. Η απόφαση είναι κοινωνική και πολιτική. Αν αποφασίσουμε να διατηρήσουμε την παραγωγή και να σας υπενθυμίσω ότι εκεί έχουμε κυρίως μικρού μεγέθους ε, εκμεταλλεύσεις, ε, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολη την επιβίωση. Ε, αν όμως επιλέξουμε να διατηρήσουμε και την παραγωγή, το ερώτημα είναι ποια μέσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε αποτελεσματικοί. Προφανώς επιδοτήσεις των επενδύσεων, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση των, ε, ε, επενδύσεων. Ε, και βέβαια χρειάζεται να ενισχυθεί οικονομικά η παραγωγή. Χρειάζονται ενισχύσεις στην παραγωγή, διότι αλλιώς η παραγωγή δεν πρόκειται ποτέ εκεί να είναι αρκετά φθηνή ώστε να επιβιώσει γνωρίζουμε ότι εκεί όλα είναι πιο ακριβά. Ε, η καλλιέργεια ε, εκταρίου εκεί χρειάζεται περισσότερο καύσιμο, χρειάζεται μεγαλύτερες δαπάνες, το οποίο σημαίνει ότι η παραγωγή είναι πιο ακριβή. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επηρεάσουμε την αγορά. Θα ήταν δύσκολο. Οπότε το καλύτερο θα ήταν να επιδοτήσουμε την παραγωγή. Αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί. Βέβαια όλα αυτά εντάσσονται και στη συνολική περιφερειακή πολιτική σε αυτές τις περιοχές. Θα πρέπει όλη αυτή η περιοχή, όλη αυτή η πολιτική να βοηθήσει τους ανθρώπους να μείνουν εκεί και να μην εγκαταλείψουν αυτές τις περιοχές. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, τώρα που έχει μοιραστεί η τράπουλα και έχει αποφασιστεί η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Οι ποσοστώσεις θα λήξουν σύντομα. Πώς όμως θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα που χρειάζονται για να επιβιώσει η παραγωγή εκεί. Ε, όλα αυτά έχουν ένα κόστος. Θα πρέπει να βρούμε τις κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης. Έχουμε ακόμα κάποια περιθώρια ελιγμών Ίσως καταφέρουμε να πείσουμε ότι είναι απαραίτητη η ε, χρηματοδότηση της παραγωγής σε αυτά τα μέρη. Κυρία Μαγκίνες, ε, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί στα σχόλια μας ό,τι αφορά τις ποσοστώσεις. Ο κύριος Χόφμαν δεν λέει ότι θα πρέπει να, ο κύριος Ντόρφμαν δεν λέει ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε τις ποσοστώσεις. Ε, απλώς σχολιάζει θέματα ισορροπίας σε αυτές τις περιοχές, τις πιο περιοχές. Ε, μην ξεχνάμε ότι αυτές οι περιοχές ε, ερημώνονται ακόμα και τώρα που υφίστανται ποσοστώσεις. Οπότε υπάρχουν και άλλα προβλήματα στις ορεινές περιοχές που ε, κατέστησαν αδύνατο οι ποσοστώσεις να κρατήσουν εκεί τον πληθυσμό. Για παράδειγμα, ε, να ρωτήσω, το 9,5% της παραγωγής του γάλατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραγόταν στις ορεινές περιοχές παλιότερα. Ισχύει αυτό ακόμα ή έχει μειωθεί. Μετά υπάρχει ένα πρόβλημα αύξηση του μέσου όρου ηλικία σε αυτές τις περιοχές, κάτι που θα δυσκόλευε την διατήρηση της παραγωγής. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς πάνε αυτοί οι παράγοντες. Και ας δούμε και τι θα προκύψει από την διάσκεψη της Κομισιόν για τον ε, τομέα του γάλατος. Ε, μετά, παράγραφοι 3, 5 και 6 έτσι και αλλιώ καλύπτονται από την μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν κάποιε επιλογέ σε ό,τι αφορά το ποιε είναι σε ό,τι αφορά το ποιε είναι οι πιο μειονεκτούσε του περιοχέ και ποιε χρειάζεται να βοηθηθούν. Ε, και να πω και το εξή. Αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό μα είναι στάσιμο και μειούμενο, θα έλεγα. Οπότε είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε όλα τα διορθωτικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της γαλακτοκομίας ε, σε αυτές τις περιοχές όταν ο προϋπολογισμός μας είναι λιτός και αυστηρός. Παρ' όλα αυτά οι προτάσεις είναι ε, ε, καλές, ε, τις καλωσορίζουμε, ε, σχετίζονται με το τι θα κάνουμε, με το τι θα κάνει η Κομισιόν το Σεπτέμβρη. Θα πρέπει να δούμε όμως και τους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που οδηγούν τον πληθυσμό των περιοχών αυτών να τις εγκαταλείψει. Όταν Πήγαμε, πήγαμε στη δική σας περιοχή κύριε Σιγητά, ε, είδαμε ότι είχαν πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις ε, και ε, που ασχολούνται αποκλειστικά με το γάλα θα είδαμε ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η παραγωγή και ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τα υπερκόστη που δημιουργεί ο χαρακτήρας της περιοχής. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ο η Κομισιόν, ο κ. Βεστέιλεν, την Γενική Διεύθυνση ε, Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο ε, Ντόφμαν για την πρωτοβουλία του και βεβαίω και συμφωνούμε ότι η παραγωγή του γάλακτο στι μειονεκτικέ, στι ορεινέ περιοχέ, στι εξόχω απόγεντρε είναι μια μεγάλη πρόκληση ε, και επίση θεωρούμε ότι η νέα ΚΑΠ δίνει κάποια εργαλεία, δίνει πεδίο ελιγμών ή στα κράτη-μέλη και την αναγκαία παραγωγή ούτως ώστε να διατηρηθεί η, η παραγωγή σε αυτές τις περιοχές. Να, παράδειγμα, κοιτάξτε, το λέει ο κύριος Ντόρμαν όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, είπαμε ότι αυτό βοηθάει με αυτή τη νέα πολιτική, ε, μειώνονται οι ιστορικές αναφορές και τα κράτη-μέλη επίσης μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν και άλλου είδους θέματα και να δουν ε, πώς μπορεί να υπάρχει η εκούσια υποστήριξη. Οπότε έτσι θα έχουμε τη βοήθεια προς αυτές τις μειονεκτικές και προς τις ε, ορεινές περιοχές. Θα πρέπει να διευρύνουμε το, τον ορισμό του τι είναι μόνιμος βοσκότυπος ή χορτολιβαδική έκταση. Οπότε έτσι να έχουμε περισσότερες ε, επιλέξιμες περιοχές που να μπορούν να είναι επιλέξιμες για αυτή την άμεση στήριξη. Και βέβαια αυτό θα πρέπει να καλύπτει την κτηνοτροφία, ε, το τοβόιο κρέας, τα πρόβατα, ε, τις αίγες. Ε, Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε σαν ανάπτυξη της πώ πώς θα έχουμε κάποιες διατάξεις που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερα προγράμματα κατά παραγγελία, δηλαδή να έχουμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες προκλήσεις, ιδίως από την γαλακτοπαραγωγή στις μειονεκτικές, στις ορεινές περιοχές και περιοχές γενικά που έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρθηκε για το πώς θα υπάρχει ειδική στήριξη όσον αφορά τις οργανώσεις των παραγωγών, κάποια δηλαδή προγράμματα για την ε, γαλακτοπαραγωγή στα όρινα, ε, επί τη βάση ε, των όσων ισχύουν για τα απορροκυπευτικά και αυτό συζητήθηκε κατά την τελευταία μεταρρύθμιση ε, οι νομοθέτες δεν θέλησαν να εκθετήσουν αυτή τη λύση διότι ιστορικά η στήριξη στα προκυπευτικά πάντοτε γινόταν μέσω των οργανώσεων παραγωγών. Όμως, όπως ξέρετε, στους γαλακτοπαραγωγούς αλλιώς γινόταν η στήριξη. Από την άλλη μεριά όμως η στήριξη για αυτό το οποίο ονομάζουμε ομάδες παραγωγών, ενώσεις παραγωγών, τώρα βάσει του δεύτερου πυλώνα είναι κάτι εφικτό για το γάλα και οπότε όλοι οι δέσμενιων μέτρων ε, τώρα υπάρχει ε, όσον αφορά ακριβώ τις οργανώσεις των παραγωγών, όσον αφορά κάποιε συμβάσει ούτω ώστε να είναι δυνατόν να αναβαθμιστούν οι πιθανότητες για τους ε, γεωργού, τους κτηνοτρόφου να μπορέσουν να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση, ευρύτερη πρόσβαση όσον αφορά την αλυσίδα της προσφοράς. έχουμε όλα αυτά. Επομένως τα μέτρα τα οποία προβλέπονται και για τις ορεινές περιοχές. Ας μην ξεχνούμε ότι σύμφωνα με την τελευταία μεταρρύθμιση έχουμε επίσης και για τις ορεινές παραγωγών διάφορες ε, δυνατότητες για το πώς θα ανταποκριθούν στις κρίσεις, της ανισορροπίες της αγοράς, ιδίω ε, όσον αφορά αυτή την περιορισμένη ε, εξαίρεση από το δίκαιο ανταγωνισμού για αυτού του είδους τις περιοχές. Εν να σας πω τώρα για αυτό που αναφέρει ο κύριος Ντόρφαμ όσον αφορά το πρόγραμμα για το γάλα στα σχολεία. Ε, αυτό το, το, το πρόγραμμα τώρα βρίσκεται υπό αναθεώρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε περαιτέρω ε, πρωτοβουλίες και έτσι να αξιοποιήσουμε περισσότερο ε, τα πλεονεκτήματα αυτού του προγράμματος και να διορθώσουμε τα μειονεκτήματα. Και ένας από τους στόχους μας είναι να δούμε πού θα βρούμε συνέργειες ε, με το πρόγραμμα για τα φρούτα στο σχολείο. Ο, αυτό είναι δόκιμο. Αυτή είναι μια πρώτη μου αντίδραση κύριε Πρόεδρε σε σχέση με αυτή την ε, έκθεση. Επίση, ε, θα είναι πάρα πολύ θετικό να συζητηθεί έτσι, να συνεχιστεί έτσι ο οργανισμό για τον τομέα του γάλακτο. Ευχαριστούμε πολύ, Παγκή ο Πρόεδρο. Και τώρα θα ξαναδώσουμε τον ε, λόγο στον εισηγητή, τον Herbert Dorfman και θα πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω τον Χέρμαν για τόσα έκανε και μας είπε όλα αυτά τα σημαντικά για αυτές τις περιοχές και φυσικά και υπάρχουν τεχνικές αλλά και πολιτικές λύσεις εις το πρόβλημα των περιοχών αυτών. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, νομίζω ότι ακόμα και η συζήτηση, η μακρά συζήτηση η οποία έλαβε χώρα και στην οποία συμμετείχαν τόσοι πολλοί συνάδελφοι και μάλιστα με καλά επιχειρήματα, καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό και από πολιτική άποψη, Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα του γάλακτος στην ε, Γεωργία. Δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα σημεία τα οποία ακούσαμε γιατί θα μακρηγορούσα υπερβολικά. Φυσικά, σύμφωνα με αυτά που είπε στην συνάδελφος Πάουλσεν για τις απόμακρες περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ παρόμοια προβλήματα με τις ορεινές περιοχές. Όλα αυτά αναφέρονται άλλωστε εκτενώς στην έκθεση. Δύο λόγια τώρα, ίσως να πω, για αυτά που είπαν οι συνάδελφοι Μποβέ και Χόσλινγκ από τους Πράσινους. Στο σημείο αυτό δεν ήθελα να ξεκινήσει μια νέα συζήτηση για τις ποσοστώσεις. Νομίζω ότι όλη η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και για τις ποσοστώσεις κατέδειξαν την πολιτική βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα στο Συμβούλιο. Ήθελα να προτείνω μέτρα τα οποία θα είναι εφαρμόσιμα. Νομίζω ότι σωστά το είπε ο συνάδελφος Άλντε, η θετική διακρατική μεταχείριση, δηλαδή αυτά τα μέτρα που δεν ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία είναι πολύ σημαντικά. Είπαν οι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη χρονική συγκυρία, γιατί έχουμε την επόμενη εβδομάδα μια σημαντική συνδιάσκεψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό και αυτό που μόνο το καταδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί και πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό και ασφαλώς δεν είναι μόνο το μοναδικό θέμα αυτό το θέμα του γάλακτος στις ορεινές περιοχές αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το είπε και η συνάδελφος το θέμα τις μεταφορές. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα αυτό, το είπε και η συνάδελφος Πάουλσεν. Είμαι πεπισμένο ότι σήμερα το υψηλότερο κόστος μεταφοράς από τις ε, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές σε ό,τι αφορά τις μεμονωμένες ε, εκμεταλλεύσεις, γιατί στους συνεταιρισμούς δεν αποτελεί πρόβλημα, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ιδιωτικές ε, τέτοιες εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση σε μία ελεύθερη αγορά αυτοί οι ιδιωτικοί αν θέλετε αγοραστές ε, θα προωθήσουν το, την πιο ευνοϊκή από άποψη κόστους ε, παραγωγή και μεταφορά γάλακτος. Αυτό θα είχε την εξή συνέπεια. Το μεταφορικό κόστος για το γάλα από ορεινές περιοχές θα ήταν ακόμα πιο ακριβό. Γιατί η μεταφορά του θα ήταν ακόμα πιο ακριβή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Ο συνάδελφο Χόισλινγκ είπε ότι τέταρτη πυλώνα δεν θα, δεν θα είναι τα κονδύλια, δεν θα μας φτάσουν τα χρήματα. Έχετε δίκιο. Είχα πει και για τον πρώτο πυλώνα όμως, είχα προωθήσει την ιδέα ενός συγκεκριμένου προγράμματος όπως είπε και η συνάδελφος Μαγκίνες, όλοι γνωρίζουμε ότι τα κονδύλια γενικά δεν πολλαπλασιάζονται. Να πω επίσης, κλείνοντας, επειδή πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι δεν μπορούμε να τα αφήσουμε όλα αυτά στα χέρια της αγοράς, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε η παραγωγή και οι μεταποιητές γάλακτος που εργάζονται σε ορεινές περιοχές τα προϊόντα τους, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και με προστατευόμενη ένδειξη προέλευσης, να μπορέσουν να συνεχίσουν να τα παράγουν και να τα διαθέτουν. Γιατί αν δεν μπορεί από μόνοι τους να τα διαθέτουν και να τα πολλούν, δεν θα μπορέσει η πολιτική από μόνη να συνεχίσει την παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές. Άρα, ναι μεν άμεση προώθηση, άμεση υποστήριξη των αγροτών στις περιοχές αυτές, αλλά και να είναι βιώσιμη η παραγωγή αυτή. Δεν συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά μπορεί να κάνουν τα κράτη-μέλη, αλλά τα μέτρα της θετικής διακριτικής μεταχείρισης σε ό,τι αφορά τις περιοχές αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν και πέρα από το 2015. Ζητώ από όλους τους συναδέλφους να μου δώσουν τα σχόλιά τους. Νομίζουν ότι αυτό που είπε και ο Μισελ Νταντά αλλά και άλλοι συνάδελφοι ότι θα πρέπει να μιλήσουμε με μια ενιαία φωνή είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα θα φροντίσω τα σχόλια που θα λάβω να τα διατυπώσω με τέτοιο τρόπο προκειμένου να υποστηρίξει το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία της Επιτροπής την έκθεση και προκειμένου να στείλουμε την έκθεση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ Χέρμπερτ και ελπίζω ότι θα υπάρχει μια ευρεία συνένεση για την έκθεσή σου. Οπότε, τώρα πάμε στο τελευταίο θέμα της σημερισίας διατάξεως. Μείνουμε το, το 9 ε, όσον αφορά την ε, διαχείριση που σχετίζεται με τι ε, δαπάνε τη τροφική αλυσίδα για ζώων, καλομεταχείριση ζώων, φυτά και αναπαραγωγικό υλικό. Τον Μάιο του 2013, σας πενθυμίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 4 από πέντε προτάσεις οι οποίε αποτελούν ε, τμήμα αυτή τη θεσμής μέτρων για την υγεία ζώων και φυτών. οπότε έτσι θα υπάρχει εφαρμογή όσον αφορά ε, κάποια, τα πρότυπα, προδιαγραφέ, υγεία και ασφάλεια όσον αφορά όλη την ε, ε, αγροτοδιατροφική αλυσίδα. Έχουμε επίσης το δίκαιο για, την, τα φυτογενομικά και επίσης ε, για την απαγωγή των φυτών όπως και την υγεία των ζώων. Έχουμε αυτή την πέμπτη πρόταση η οποία εγκρίθηκε τον Ιούνιο και αυτό αποτελεί το, θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Καλύπτουμε τις οικονομικές πλευρές αυτού του νομοθετικού πακέτου, αλλά επίσης και τη δαπάνη, τους πόρους που έχουν δεσμευτεί για τα διατροφή αλλά και, τα, και την τροφή των διατροφικών ζώων τις 14-2020 και όλα αυτά θα συνεχίσουν πρώτα από το 2014 οπότε και εμείς θα πληρώσουμε τις για το ζήτημα πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση για το υπόλοιπο πακέτο μέτρων. Οπότε και θες αμέσω να δώσω το λόγο στην συνάδελφο Ανιές Λεμπράν. Ευχαριστώ πολύ. Ο, ο είπε ότι αυτός ο κανονισμός αποτελεί τίμα του πακέτου που δημοσιεύθηκε, δόθηκε στη δημοσιότητα, δημοσιότητα στις 6 Μαΐου. Περιλαμβάνει πέντε κείμενα αυτού του πακέτου, τέσσερα ε, τομεακά και τον κανονισμό διαχείρισης των, δαπανών που έχει ως στόχο να απλοποιήσει το νομοθετικό πλαίσιο που έχει σχέση με την διατροφική αλυσίδα. Στο πλαίσιο αυτής της απλοποίησης θα καταργήσει και θα τροποποιήσει 11 παλαιότερες νομικές πράξεις. Το είπατε και εσείς Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει να υιοθετηθεί σε πρώτη ανάγνωση και γι' αυτό το λόγο είναι χρήσιμο να εργαστούμε ε, γρήγορα στις 25 Νοεμβρίου θα πρέπει να υιοθετηθεί στην Επιτροπή έκθεση έτσι ώστε να μεσολαβήσει ε, αρχές του επόμενου χρόνου ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, η αρχική έκδοση του, εκδοχή του χρονοδιαγράμματος μάλιστα δεν επέτρεπε την σημερινή συζήτηση. Ορισμένες ε, από τις διατάξεις υπάρχουν ήδη, αλλά υπάρχουν και τρεις καινούργιες. Πρώτον, εκλογήκευση, εξορθολογισμός ε, των ε, ποσοστών συγχρηματοδότησης. Έχουμε τρία ποσοστά αυτή τη στιγμή. Ένα μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 50%, ένα μέγιστο ποσοστό κατεξαίρεση του 75% για τις διαμεθοριακές δράσεις μεταξύ κρατών μελών, τουλάχιστον δύο κρατών μελών και για τα κράτη-μέλη που έχουν ε, κατακεφαλήνα ΑΕΠ κάτω του 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά έχουμε ένα τρίτο ιδιαίτερο μέγιστο ποσοστό 100% για την περίπτωση φυτογενομικών κινδύνων, μεγάλων φυτογενομικών κινδύνων ε, ή για δράσεις ε, που λαμβάνουν χώρα από και σε τρίτες χώρες. Έχουμε ένα κατόφλι 50.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε κάτω από το οποίο δεν είναι δυνατόν να δοθεί ε, επιδότηση. Παλιότερα δεν υπήρχε κατόφλι. Όμως, ε, εντάξει, φανταζόμαστε του λόγους. Ε, δεύτερο καινούριο στοιχείο έχει σχέση με την δημιουργία δικτών. Ε, οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή δεν την χάνουν κατάλληλη αξιολόγηση. Οπότε η Κομισιόν προτείνει τη δημιουργία συγκεκριμένων δικτών για να αξιολογούμε καλύτερα τα αποτελέσματα των πολιτικών μας στην διατροφική αλυσίδα. Τρίτο καινοτόμο στοιχείο αφορά τα προγράμματα έρευνας και προγράμματα παρακολούθησης βλαβερών οργανισμών προκειμένου να προλάβουμε κινδύνους στην ε, φυτική παραγωγή. Αυτά είναι τα βασικά καινούρια σημεία που προσφέρει το κείμενο. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω δύο σημεία. αυτό που μόλις είπα προηγουμένως, αλλά και ένα δεύτερο θέμα, το θέμα των πράξεων κατά εξουσιοδότηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τον κατάλογο ασθενειών. Θα πρέπει να δούμε την κατανομή ανάμεσα στις ε, βασικές πράξεις, πράξεις ε, ε και τις εκτελεστικές πράξεις και επίσης να δούμε το θέμα του αποθεματικού κρίσης και της πρόσβασής του σε αυτό. Αυτά προς στιγμή. Ε, προς το παρόν θέλω να ακούσω τα σχόλιά σας, να καταγράψω τις ερωτήσεις σας και ενδεχομένως να δώσω και κάποιες απαντήσεις μετά τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Η κυρία Γαρθία Πέρεθ καταρχήν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Λεμπρά για την πρώτη αυτή παρουσίαση των ε, τροποποιήσεων που φέρνει η Κομισιόν μέσω αυτού του κανονισμού. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά προκειμένου να υποβάλουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις, ε, προτάσεις τροποποίησης του κειμένου. Σε αυτή την πρώτη συζήτηση θα κάνω κάποια γενικά μόνο σχόλια ε, που εστιάζουν σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, η πρόταση προβλέπει μείωση κατά 30% των ε, πόρων σε σχέση με την, ε, περίοδο, την τρέχουσα περίοδο. Ε, θεωρώ ότι στην περίπτωση που θα χρειαστούν περισσότερα κονδύλια θα πρέπει να διαθέτουμε και άλλους μηχανισμούς πέραν του αποθεματικού κρίσης που να έρχονται από τον τομέα 3 ή από άλλους τομείς του προϋπολογισμού εφαρμόζοντας την αρχή της ευελιξίας. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε υπάρχει περίπτωση να ε, ε, πυροδοτηθεί ο μηχανισμός της δημοσιονομικής πειθαρχίας τον οποίο από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να εφαρμόζουμε ετησίως. Εμείς ως Επιτροπή είχαμε εκφράσει και στο παρελθόν μας τις ανησυχίες μας για τον μηχανισμό δημοσιονομικής ε, ε, αυστηρότητας, ε, πειθαρχίας. Ιδιαίτερα όμως για αυτό τον τομέα, ιδιαίτερα για αυτό μάλλον το, το κείμενο, για αυτό το κομμάτι θα πρέπει να βρούμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες υποβολής των εκθέσεων τις προθεσμίες. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστική πρόταση Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται πριν από τις 31 Μαρτίου να υποβάλουν ε, λεπτομερή τεχνική έκθεση για το προηγούμενο έτος. Ε, η προθεσμία αυτή είναι πολύ στενή, ιδιαίτερα για ορισμένες χώρες όπως ενδεχομένως η δική μου που η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες από τις αυτόνομες περιοχές μας που έχουν τις την αρμοδιότητα κατά τόπους. Οπότε πιστεύω ότι η προθεσμία θα πρέπει να είναι 30 Απριλίου όπως σήμερα. Σε ό,τι αφορά την, τον κατάλογο των ασθενειών, ε, ε θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος βάσης και η Κομισιόν απλώς να προσθέτει να φέρει όχι όλα να αποφύονται στην Κομισιόν με εκτελεστική πράξη. Μετά, το κατόφλιτο 50.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων ε, αφήνει απ' έξω χώρες που έχουν ε, μικρές ανάγκες αλλά για ασθένειες που μπορεί να είναι πολύ σημαντικές κατά τα άλλα. Αυτές είναι Αυτά είναι τέσσερα θέματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να τα δει η Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε λέει ο Οπότε τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Κύριε Φαν Γκέρτον. Ναι, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Σας ευχαριστώ γιατί τόσο διεκπαιρεωτικά χειριστήκατε αυτή την πρόταση. Όπως προείπατε, είναι πολύ σημαντικό αυτή η πρόταση να εγκριθεί ε, όσο γίνεται ε, πιο γρήγορα ε, ή δυνατόν πρώτο τέλος του έτους. Όπως εξήγησε η συγγήτρια, η πρόταση αυτή κωδικοποιεί την υπάρχουσα νομοθεσία, να είναι πιο εύκολο τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν νομοθεσία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης. Καλύπτει όλες τις δαπάνες όσον αφορά τη διατροφή και τη, τη, την τροφή των ζώων. Είπαμε ότι έχουμε και τα θέματα της γρήπης στην Ιταλία. Έχουμε επίσης τα εργαστήρια αναφοράς όπως για τις διοξίνες και για τα τροποποιημένα στους οργανισμούς όλα αυτά προβλέπονται, συνδέονται με την πρόταση όλα αυτά είναι τμήμα αυτού του πακέτου μέτρων και έτσι θέλουμε να υπάρχει ένα κέντρο αναφοράς για την καλοπτυχία των ζώων, που βλέπετε ότι καλύπτουμε μια ευρεία γκάμα από δραστηριότητε όσον αφορά κτηνοτροφέ και διατροφή. Επίση, ανέφερε η κυρία Πέρεθ ότι συρρυκνώθηκε η πρικοδότηση. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αλήθεια. Είναι περίπου το ίδιο όπως και πέρσι. 262 εκατομμύρια, ακριβώς όσα προβλέπονται ε, και φέτος θα είναι και του χρόνου, θα είναι και του χρόνου, θα είναι και πέρσι, άρα δηλαδή δεν έχουμε μειώσει ε, την πρικοδότηση. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι ε, επειδή έχουμε την βουκέλωση, επειδή έχουμε την, την φυματίωση, έπρεπε να λάβουμε δράση την τελευταία δεκαετία, οπότε και είπαμε να μην μειωθεί ο Προπολογισμό. μη όχι μάλλον για, για τέτοιου δράσεις, αλλά όχι ο γενικό προπολογισμό και έχουμε 1,8 δις για τελευταία επταετία. Η κυρία Πέρεθ και η συγγήτρια αναφέρανε το θέμα της προσβασιμότητας ε, στα, στο αποθεματικό του προπολογισμού. Όπως ξέρετε αυτό ήταν ε, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν πριν το Σάμερ. Οπότε και εγκρίθηκε ο προπολογισμός για την ε, ΚΑΠ. Με τους λόγους αυτό δεν μπήκε στο τελοκείμενο, πάντως ε, ο Επίτροπος όλος ήταν ε, σαφής και σας έγραψε σε σχέση με την τροποποίηση του παλαιού άρθρου 4ε. το περιεχόμενο αυτό τώρα προκαλείται το άρθρο 5. Πολλές φορές έχουμε τεράστιες κρίσει όλοι θα θυμάστε ε, τον αυτό πυρετό το 2001 στο Βασίλειο θυμάστε τι έγινε με την ασθένεια εκείνη της μπλε Indeed, the budget which is foreseen is not enough. Και για αυτό το λόγο η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ε, καλύπτει κάποιες ε, εξαιρετικές περιστάσεις σύμφωνα με τις οποίες καλύπτονται πρικοδοτούνται ε, οι αντιμετωπίσει αυτών των κρίσεων και πέρεθε επίση τώρα ανέφερε τι διάφορε καταληκτικέ ημερομηνίε. Μα είπε Μάρτιο σε σχέση με Απρίλιο τι προτιμάει. Αυτό πάντω συνδέεται και με του δείκτε που αναφέρθησαν από την κυρία Λεμπρά. Εμεί αυτό το οποίο θέλουμε είναι έχουμε έχουν περίπου λίγο λιγότερο από 200 εκατομμύρια. Και θέλουμε αυτά τα χρήματα να πιάνουν τόπο. Οπότε τώρα αυτό το οποίο θέλουμε, αυτή η έκθεση να είναι έτοιμη τον Μάρτιο του χρόνου. Θέλουμε το πρόγραμμα να είναι αποτελεσματικό, ελσχεσικό στους αποτελέσματος. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια ευελιξή σχέση με αυτό το Μάρτιο-Απρίλιο όσον αφορά την έγκριση του προγράμματο. Κάτι άλλο, το τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε είναι τα 50 εκατομμύρια σαν όριο για το πρόγραμμα. Και αυτό αντικατοπτρίζει τη θέση μας όσον αφορά το διοικητικό άρθρο, αλλά μέχρι σήμερα η πρόταση τη επιτροπή ήταν το πρόγραμμα αυτό να μην ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, όχι, αν, αλλιώς δεν θα το η Ένωση. Ξέρετε βέβαια ότι έχουμε κάποια μικρά, πολύ μικρά μέλη, πολύ μικρά προγράμματα που εκεί επιβάλλεται η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και αν το κόστος είναι κάτω από 50 εκατομμύρια. 50.000. Άρα και από πλευρά μα πρέπει να επιδείξουμε κάποια ευελιξία. Σα ευχαριστώ. Και επίση ελπίζω το συντομότερο δυνατόν να εγκριθεί η έκθεση. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα ξαναδούμε στο λόγο στην κυρία Λέμπρα. Ευχαριστώ για αυτές τις παρατηρήσεις. Αυτά που, είπαν, που είπε η κυρία Γκαρσία Πέρε, ε, νομίζω ότι είναι προσωστή σωστή κατεύθυνση ε, σύμφωνα με αυτά που είπα εγώ σε ό,τι δεν η Κομισιόν ε, βλέπω ότι συμφωνεί με την ευελιξία σε ό,τι φοράει το χρονοδιάγραμμα σε ό,τι φοράει το κατόφλι αν κατάλαβα καλά η Κομισιόν λέει πω είναι τόσε λίγε οι παρεμβάσεις, κάτω από 50.000 που αξίζει το λόγο να έχουμε ένα ελάχιστο. Απ' την άλλη μεριά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επιχείρημα ακριβώ αντίστροφα. Επειδή ακριβώ είναι πολύ λίγε οι επεμβάσει ε, που γίνονται για ποσά κάτω 50.000 ευρώ, γιατί να βάλουμε κατόφλι, αφού έτσι και δεν θα αλλάξει τίποτα. Για τον κατάλογο των ασθενειών, όπως ε, είπα και εγώ στην αρχή, νομίζω ότι η κυρία Γκαρσιά ε, ε, έκανε τη σωστή παρατήρηση και ότι δεν αφορά το θέμα του αποθεματικού κρίσεων. Η Κομισιόν πολύ σωστά αναφέρει ότι χάρη στις δράσεις επαχρήμησης και παρακολούθησης μπορούμε να ελπίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει να αντιμετωπίσει όλο και λιγότερα ε, οδυνηρά περιστατικά ασθενειών στο μέλλον. Όμως, παρόλο ότι έχουμε πραγματική μείωση τέτοιων κρουσμάτων σε ό,τι αφορά την υγεία των ζώων, αντιθέτως έχουμε αύξηση στις ασθένειες και στα περιστατικά που συμπεριλαμβάνουν φυτά. Οπότε ε, ας μην βιαστούμε να πανηγυρίσουμε. Ασφαλώς θα πρέπει να εμπιστευτούμε τα μέτρα που λαμβάνουμε, αλλά να έχουμε και στο μυαλό μας ότι υπάρχει περίπτωση στον φυτο-υγειονομικό τομέα να έχουμε περίπλοκες καταστάσεις στο μέλλον. Αυτά και θα επανέλθουμε με καινούργια στοιχεία σε μια επόμενη συνάντηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο τις εργασίες μας ε, σήμερα. Η υποβολή της έκθεσης κ. Λεμπρά θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, τροπολογίες μέχρι τις 20 Οκτωβρίου και θα ψηφίσουμε στις 25 Νοεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας υπενθυμίζω ότι αμέσως μετά έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών μαζί με τους κοιόδης ηγητές για τα, τις τελευταίες διαπραγματεύσεις για την ΚΑΠ. Ένα τέταρτο διακοπή και μετά ξεκινάμε τη σημαντική αυτή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας.